Good afternoon, colleagues. Thank you for being here. Καλημέρα σας, λέει ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος Μωράης δεν θα είναι εδώ σήμερα το απόγευμα, οπότε θα προεδρεύσω εγώ σήμερα το απόγευμα της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Το πρώτο μας θέμα, ως συνήθως, είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ε, ε, και έχουμε την εξή μεταβολή, το σημείο 12 όσον αφορά την παρουσία του σχεδίου έκθεση για ανταλλαγή, συνδρομή και κατάρτιση όσον αφορά το πρόγραμμα προστασία του ευρώ για παραχάριξη και ευδηλία 2021 με 27 περίκλη 4 το εν λόγω σημείο λέγω αναβάλλεται. Ελπίζω να υπάρχει κάποια ένσταση σε αυτό που σας ανέφερα οπότε εγκρίνεται η μερίσια διάταξη και προχωρούμε τώρα Εστά της διερμηνίας σήμερα. Έχουμε σε όλες τις γλώσσες, μάλλον από όλες τις διερμηνία, εκτός από τα κελτικά και αύριο θα έχουμε πάλι όλες τις γλώσσες εκτός κελτικών, κροατικών και μαλτέζικων. Και τώρα, όσον αφορά την έγκριση των προτάσεων των συντονιστών, ε, σύμφωνα με το άρθρο 205. Έχουμε το σημείωμα των συντονιστών σε σχέση με την έγγραφη διαδικασία της 19ης ενδεκάτου του 18 και τον ορισμό εισηγητών. Ο Κλοντ Μοράς, ως πρόεδρος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, ορίστηκε εισηγητής για το σχέδιο κανονισμού που τροποποιεί τον κανονισμό του Συμβουλίου 539 του 2001, όπου ε, απαριθμούνται οι τρίτες χώρες των οποίων οι υπήκοοι θα πρέπει να κατέχουν θεωρήσεις διαβατηρίων, ότι είναι σύνορα τα εξωτερικά σύνορα κλπ. Σε σχέση και με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Σοφία Νετφέλντ είναι η συγγήτρια για το ψήφισμα όσον αφορά τι δραστηριότητε ομάδα εργασία με την γενική εντολή για καταπολέμηση τη ε, διαφθορά ε, του κράτου δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένε περιπτώσει όπω ε, Μάλτα και Σλοβακία. Ο υποφαινόμενο ορίστηκα ο εισηγητή μα όσον αφορά την έκθεση τη πρωτοβουλία για τι ανθρωπιστικέ θεωρήσει. Και έχουμε την ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων ε, Αφρικανική καταγωγή στην Ευρώπη. Και έχουμε την απόφαση των συντονιστών τη 27 Ενάτου του 18, οπότε και δεσμευτήκαμε να προετοιμάσουμε ένα σχέδιο ε, όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα αυτών των ανθρώπων και συμφωνήσαμε οι πολιτικέ ομάδε να ε, προτάξουμε, να διατυπώσουμε μια προφορική ερώτηση προ την Επιτροπή και αυτό θα υποβληθεί στην διάσκεψη των Προέδρων, ούτω ώστε να καλυφθεί, να ενταχθεί στη μέση διάταξη τη Συνόδου του Ιανουαρίου με συζήτηση. Και θα συμπληρωθεί διαδικασία με ψήφισμα σύμφωνα με την διάταξη 168 παράγραφος 5. Αυτές οι προτάσεις των συντονιστών και ελπίζω ότι εγκρίνονται από την Επιτροπή χωρίς ενστάσεις. Παρακαλώ. Όσον αφορά τις ε, και εφαρμοστικέ πράξεις, έχουμε μία ανακοίνωση που αφορά την 7η αποφάση όσον αφορά το συστημα εισοδου εσόδου-εξόδου και το σχετικό κανονισμό. Ε, πρόταση κάποια έγγραφα και αφορούν ένα σύστημα αδειοδότησης, το σύστημα αιτιάς και επίσης έχει κάποιες ε, τεχνικές λύσεις όσον αφορά το σημείο πρόσβασης προς το σύστημα αιτιάς και ε, έτσι να διευκολυνθεί η συλλογή δεδομένων από την Ένωση και από την Europol. Επίσης έχουμε την απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την χρήση των ε, ε, δακτυλικών αποτυπωμάτων για αυτό το σύστημα εισόδου-εξόδου και εδώ αναφέρονται οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις για αυτό το σύστημα εισόδου-εξόδου και αναφέρονται οι προϋποθέσεις και τα μέτρα για την διαλειτουργικότητα μεταξύ του συστήματος εισόδου-εξόδου και του συστήματος πληροφοριών θεωρήσεων διαβατηρίου. Η βασική νομοθετική πράξη είναι ο κανονισμός 2017-22-26 που θα σπίζει αυτό το σύστημα εισόδου-εξόδου για αυτά τα ε, δεδομένα όσον αφορά υπηκός τρίτων χωρών. Εκεί οριζόνται οι προϋποθέσεις πρόσβασης στο σύστημα εισόδου-εξόδου και τροποποιείται η σύμβαση που εφαρμόζει την συνθήκη του Σέγγεν και τους κανονισμούς 767 ε, και 1077. Η παραλαβή αυτής της εφαρμογής πράξης κοινοποιήθηκε σε όλους τους συναδέλφους της ΛΥΜΠΕ και έχουμε το newsletter, το ενημερωτικό δελτίο μας, στις 23 η ενδεκάτου που αναφέρονται όλα αυτά. Αν θέλετε να βγάλετε κάποια ένσταση, παρακαλώ ενημερώστε την γραμματεία μας πριν τι 4 το μεσημέρι. Η ηλεκτρονική ψηφορία θα γίνει αύριο στις 9 και 4. Οπότε, να είστε σίγουροι ότι δεν ξεχάσατε την ε, ηλεκτρονική σας κάρτα για την ψηφοφορία. Να δούμε τώρα τα σήμερα της διατάξεως. Έχουμε το σημείο υπαριθμών 3. Αξιολόγηση του κινδύνου του οργανωμένου εγκλήματος στο διαδίκτυο. Προβλέπεται παρουσίαση από τον κύριο Φίλιπ Αμάν, ο οποίος είναι τμήματάρχης στρατηγικής στο κέντρο κυβερνοεγκλήματος της ε, Europol. και ξεκινούμε αυτή την παρουσίαση όσον αφορά την ε, αξιολόγηση του κινδύνου του 2018 και ε, εδώ έχουμε ε, τα θέματα της δραστηριότητα της Europol όσον αφορά την ανάλυση των αδειωμένων απειλών και των πιο βασικών εξελίξεων όσον αφορά το κυβερνό έγκλημα πέρσι και τις βασικές τάσεις και εξελίξεις και επίσης θα μας διατυπώσει κάποιες συστάσεις, θα του δώσω το λόγο του κύριου Αμάν και κατόπιν ε, έχουμε ερώτα απαντήσει από τους συναδέλφους. Κύριε Αμάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την ευκαιρία που μας δίνετε να σας παρουσιάσουμε την ετήσια αξιολόγηση απειλής του οργανωμένου εγκλήματος στο διαδίκτυο. Ε, είναι μια έκθεση που εδώ και πέντε χρόνια δημοσιεύουμε ετησίω. Όπως είπατε, είναι μοναδική αυτή η αξιολόγηση, γιατί επικεντρωνόμενοι στο, στο όργανο επιβολής και στι αρχέ επιβολή του νόμου, δίνουμε πληροφορίες ε, με συμμετοχή του κλάδου, των πανεπιστημίων και δίνουμε πληροφορίες ε, για τους, ε, τις απειλές, τις τάσεις στον κυβερνοχώρο, ενημερώνουμε για τις προτεραιότητες και παρέχουμε και συστάσεις ενημερώνοντας τους δίνοντες πολιτικής και τα αρχές επιβολής του νόμου και ενημερώνουμε και τους πολιτικούς, τους δίνοντες για τη λήψη αποφάσεων ε, για να τεκμηρώσει τις αποφάσεις τους σε πολλούς τομείς. Σε ό,τι αφορά την φετινή μας έκθεση, καταρχήν ε, οι εταίροι μας από τις ε, αρχές επιβολής του νόμου από τα κράτη-μέλη μας στέλνουν τις ερευνές τους. Έχουμε έρευνες τρίτων μερών, συμβουλευτικών ομάδων. Έχουμε ένα για το ίντερνετ, για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και για τους παρέχοντες ε, υπηρεσίες επικοινωνίας, στηρίζει τέτοιες ε, συμβουλευτικές ομάδες και επίσης και έρευνα από δημόσιες πηγές. Πάμε στην επόμενη διαφάνεια, καλύπτοντας ε, ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και επικεντρωνόμαστε κυρίως σε τρεις γιατί το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Κλίματα στον κυβερνοχώρο βρίσκεται στο κέντρο επιχειρήσεων της Europol και ασχολείται με απάτες πληρωμών, καταπολέμηση παιδικής προνογραφίας στο διαδίκτυο ε, και διάφορες άλλες μορφές ηλεκτρονικής απάτης. Επίσης, ε, εξετάζουμε ακόμη και κβαντική, υπολογιστική, συναφή δηλαδή θέματα. Και αν δούμε ένα χρόνο πριν και ποιες ήταν βασικές εξελίξεις ε, και οι τάσεις, ε, προσπαθούμε με βάση αυτά τα στοιχεία να προβλέψουμε τις τάσεις και το μέλλον για τον επόμενο χρόνο, το επόμενο δωδεκάμενο. Ποιες ήταν ε, οι βασικές εξέλιξεις. Καταρχήν, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας των Δεδομένων μαζί με την Οδηγία για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ήταν τα βασικά νομοθετικά στοιχεία για την ασφάλεια στον χώρο και τα χρησιμοποιούμε και εμείς αυτά τα δύο μέσα, το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και την Οδηγία για να αυξήσουμε το σενάριό μας για την ασφάλεια, για τις αρχές επιβολής του νόμου, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις με την αύξηση της παράβασης της εξαγωγής ή αντιγραφής δεδομένων και προσπαθούμε να διαρευνήσουμε τέτοιου είδους ε, παραβάσει στο διαδίκτυο για εξαγωγή και αντιγραφή δεδομένα είχαμε μια πολύ επιτυχημένη συντονισμένη δράση για να αντιμετωπίσουμε τις εγκληματικές δραστηριότητες του Darknet, του σκοτεινού διαδικτύου. Κλείσαμε τις ε, δύο μεγαλύτερες ε, αγορές που ήταν το Alphabay και η Χάνσα και στο μεταξύ και μια τρίτη το Ramp και άλλο σημαντικό θέμα είναι το γεγονός ότι τα κρυπτονεμίσματα γίνονται πλέον κάτι το συνηθισμένο γιατί είναι ένας θεμητός ε, τρόπος πληρωμής και τα κρυπτονομίσματα. Αλλά ακριβώς επειδή είχαμε μια έξαρση, ε, αύξηση της αξίας, της αξίας των κρυπτονομισμάτων, έγιναν και αυτά ε, στόχαστρο των εγκληματιών στον κυβερνοχώρο. Σε ό,τι αφορά τις ε, τάσεις και τις απειλές, σίγουρα το λιτρισμικό, το κακόβουλο λογισμικό ransomware, ε, λιτρισμικό δηλαδή, είναι από τις βασικές απειλές, εξακολουθεί να κυριαρχεί. Αν λάβουμε υπόψη και το crypto jacking, δηλαδή πειρατεία υπολογιστών που χρησιμοποιούνται από εγκληματίε ε, για να χρησιμοποιηθεί η επεξεργαστική ισχύ του υπολογιστή σας για να κάνουν mining, εξόρευση δηλαδή κρυπτονομισμάτων. Αυτή είναι μια νέα τάση, το cryptojacking, που μάλιστα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και χωρίς πολύ κίνδυνο είναι μια πηγή εισοδήματος ε, για τους ε, παραβάτες. Επίσης έχουμε ε, παράνομη αγορά που προσφέρει εξοπλισμό και εξαρτήματα για την κατανεμημένη επίθεση άρνης εξυπηρέτησης, επιθέσεις DDoS όπως λέγονται. Και δυστυχώς υπάρχουν εξοπλισμοί που μέσω σε ένα μήνα και χωρίς ιδιαίτερη τεχνογνωσία μπορείτε να νοικιάσετε τέτοιες υπηρεσίες και τέτοιο εργαλεία και να προβείτε σε επίθεση άνεσης εξυπηρέτησης. Τα κίνητρα αυτών που τη διαθέτουν είναι πολιτικά, οικονομικά, ε, πάντως χρησιμοποιούνται σε αυτές τις παράνομες αγορές ε, και διατίθενται τέτοια εργαλεία. Επίσης, ε, Έχουμε πολλές ηλεκτρονικές απάτες με τις κάρτες Card Not Present, CNP. Είναι πολύ χαρακτηριστικές τέτοιες ε, οι κάρτες. Γίνεται κλωνοποίηση αυτών των καρτών και πληρώνονται σε άλλες χώρες ε, χρηματικά ποσά. Και επίσης, ε, επειδή είχα αύξηση της αξίας του bitcoin και άλλων κρυπτονομισμάτων, πέρυσι ένα bitcoin ήταν 19.000 δολάρια και γι' αυτό έγιναν ε, στόχος ε, οι ιδιοκτήτες ε, κρυπτοπορτοφολιών πορτοφολιών ή ανταλλάκτες τέτοιων κρυπτονομισμάτων έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των παραβατών. Επίσης και παιδική πορνογραφία είναι σημαντικό θέμα. Πολλές φορές παρακάμπτονται τεχνητοί έλεγχοι και σίγουρα το διαδίκτυο, το darknet, ε, δημιουργεί τεράστιες απειλές και για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, αλλά και για συμβατικού είδους εγκλήματα. Αλλά έχουμε και παιδική εκμετάλλευση και κακοποίηση, παιδική πορνογραφία και είχαμε αύξηση της παιδικής πορνογραφίας και αύξηση και των εργαλείων επικοινωνίας για τη διανομή τέτοιου υλικού παιδικής πορνογραφίας θα δούμε τώρα πιο λεπτομεριακά αυτές, αυτούς τους έξι τομείς. Καταρχήν, έγκλημα που εξαρτάται από τον κυβερνοχώρο. Είναι κάποιες αξιόπινε πράξεις που υπάρχουν ακριβώ επειδή έχουμε το διαδίκτυο. Χωρί το διαδίκτυο δεν θα ήταν, δυνατάτε, δεν θα ήταν δυνατή διάπραξη τέτοιων εγκλημάτων. Το λιτρισμικό είναι βασική απειλή, σπαμ, ε, αλλά θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην πρόληψη και στην επαγρύπνηση. Επίσης, ε, έχουμε διάφορες μορφές επίθεσης, την κοινωνική μηχανική χειραγώγηση, δηλαδή spam και email που μολύνουν οι υπολογιστές. Και επίσης έχουμε και αυτή την ε, πειρατεία για mining κρυπτονομισμάτων, το cryptojacking, που έχει γίνει ένα πολύ δημοφιλές μέσο για τους εγκληματίες ε, για να βγάλουν χρήματα. Κάτι που παρατηρούμε επίσης είναι σε κάποιες, ότι σε κάποιες γεωγραφικές ζώνες και με βάση τα στοιχεία που έχουμε λάβει, στη Δυτική Αφρική έχουμε πολλούς παραβάτες που μετατοπίζονται προς τον κυβερνοχώρο και επιτίθενται κατά ευρωπαϊκών υποδομών κυρίως. Και επίσης έχουμε αύξηση των επιθέσεων ε, των ιδιοκτητών κρυπτονομισμάτων ή ε, πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων ή ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων. Έχουμε ένα κεφάλαιο που αφορά τη σύγκληση του κυβερνοεγκλήματος και της τρομοκρατίας. Βλέπουμε ποιες είναι οι κυβερνοεγκανότητες των τρομοκρατών στον κυβερνοχώρο και κάνουμε μια επισκόπηση των διαφόρων εξελίξεων που έλαβα χώρα το τελευταίο ε, με ιδιαίτερη εστίαση στην ε, κύβερνο διάσταση και εξετάζουμε κυρίως ε, το Ισλαμικό κράτος που ήταν πολύ αποτελεσματικό σε ό,τι φορά τη χρήση του διαδικτύου για την ε, διανομή της προπαγάνδας, αλλά έχουν και άλλοι υπόλοιπες κυβερνοικανότητες του Ισλαμικού κράτους, θα μάλλον περιορισμένες. Επίσης, χάρη σε αποτελεσματικές δράσεις μας όπως είναι το κλείσιμο του Χάρσε και του Αλφαμπέι περιορίσαμε τις δραστηριότητες στο σκοτεινό διαδίκτυο, το Darknet. Έτσι έχουμε αλλαγή κάποιων διάβλων, μετακίνηση προς πιο μικρές αγορές, οπότε σίγουρα το κλείσιμο αυτών των τριών βασικών αγορών επηρέασε. Σε ό,τι αφορά τις αξιόπινες δραστηριότητε του σκοτεινού διαδικτύου έχουμε ένα κατακαιρματισμό και κυρίως λαθρεμπόριο ναρκωτικών που επικρατεί σε αγορές του σκοτεινού διαδικτύου. Άλλη σημαντική απειλή είναι, όπως σας είπα, οι απάτες πληρωμών. Ακριβώς το λόγο του ρόλου του Europay, του, της Mastercard και της Visa. Έτσι έχουμε πολλές απειλές με κάρτε κάρτες πληρωμών και οι πληρωμέ δεν γίνονται στην Ευρώπη. Είναι καλή οργάνωσή του, γιατί κλωνοποιούνται οι κάρτες στην Ευρώπη, αλλά οι πληρωμές γίνονται σε εξωκοινωτικές χώρες, οπότε τα χρήματα μπορούν κάποια στιγμή να επιστρέψουν σε οργανωμένο έγκλημα που βρίσκεται στην Ευρώπη. Επίσης έχουμε ειδικέ ε, επιθέσει κατά ATM και κατά POS, κατά σημεία, πόλη, κατά Επίσης έχουμε κάποιε εικονικέ εταιρείε. Ε, που χρησιμοποιούν την απάτη μέσω τηλεπικοινωνιών, που είναι ανερχόμενη απειλή και δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις στις αρχές επιβολής του νόμου. Ιδιαίτερα στο θέμα της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο βλέπουμε τους δράστες που είναι πολύ αποτελεσματικοί σε ό,τι αφορά τα, τα πρότυπα και χρησιμοποιούν την κρυπτογράφηση, το TOR, το Tor είναι μια απόλυτα νόμιμη πλατφόρμα, αλλά γίνεται αξιόπινη χρήση της, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα στις αρχές επιβολής του νόμου. Έτσι, οι έρευνες ε, των ομάδων αυτών διακίνηση παιδικής πορογραφία είναι πολύ δυσχερείς λόγω τη χρήση τέτοιων ε, μεθόδων κρυπτογράφηση του TOR. Επίσης χρησιμοποιούνται και άλλες ε, εμπορικέ πλατφόρμες επικοινωνίας για τη διανομή υλικού παιδικής προγραφίας. Επίση, χρησιμοποιείται η κρυπτογράφηση κάτι που δημιουργεί πρόβλημα στις αρχές επιβολής του νόμου. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, δεν επισημαίνουμε τις τάσεις και τις απειλές, αλλά προβαίνουμε και σε κάποιες συστάσεις για τις αρχές επιβολής του νόμου, ενημερώνουμε τους ηθήνοντες για τη λήψη αποφάσεων και κάνουμε συστάσεις στους εταίρους μας από τον κλάδο. Χρειαζόμαστε πάντως ένα δίκτυο συνεργασίας για να καταπολεμήσουμε αυτά τα εγκληματικά κυκλώματα και είναι σημαντικό όλοι οι εμπλεκόμενοι να, όλοι οι εμπλεκόμενοι να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους στα πλαίσια φυσικά τα νομικά. Σε ό,τι αφορά τη, τους κυβερνοεγκληματίες έχουμε αφενός ε, κάποια εγκλήματα χαμηλής αξίας ε, υψηλού όγκου εμείς ε, επικεντρώμαστε κυρίως στην πρόληψη σε ό,τι αφορά και την επαγρύπνηση για την κυβερνό ε, ασφάλεια, ενώ οι αρχές επιβολής του νόμου ενδιαφέρονται για τους στόχους υψηλών αξιών, ώστε να μπορέσουν να επηράσουν με ενέργειες παρέμβασης ε, την, το σκοτεινό διαδίκτυο και τις παράνομες αγορές. Και εδώ είναι σημαντικό να ευθυγραμμίσουμε όλους τους εταίρους μας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συνεργασία, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της κατάχρησης του σκοτεινού διαδικτύου. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να παρακολουθούμε τις αναδυόμενες τεχνολογίες και να δούμε πώς μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και εμείς αποτελεσματικά για να εξασφαλίσουμε καλύτερη πρόληψη, επαγρύπνηση και πιο αποτελεσματικές έρευνες. Και τέλος, εξαιτίας ακριβώς γεγονότος ότι τα κρυπτονομίσματα γίνονται πλέον κάτι συνηθισμένο, θα πρέπει να αναβαθμίσουμε και εμείς τις ικανότητές μας ε, ε, και τη τεχνογνωσία μας και εμείς και οι αρχές επιβολής του νόμου και για τα κρυπτονομίσματα. Βέβαια δεν είναι όλα ζωφερά και αρνητικά, γιατί υπάρχουν και πολλά, ε, πολλά θετικά παραδείγματα, πολλές επιτυχίες μετά από συνεργασία μας με τις ομάδες επιβολής του νόμου. Είχαμε πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις, καλή συνεργασία με τον κλάδο και είχαμε κάποιες εκστρατείες επαγρύπνησης και πρόληψης. Βλέπετε εδώ πολύ άριθμα παραδείγματα τέτοια συνεργασία. Οπότε μπορούμε να είμαστε κάπως υπερήφανοι, αλλά σίγουρα θα πρέπει να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας, γιατί είναι ραγδαία η εξέλιξη των τεχνολογιών και θα πρέπει να είμαστε πιο προαιρετικοί και να μας ξεπερνούν οι εξέλιξεις. Θα πρέπει να συνεχιστεί η υπάρχουσα συνεργασία και να αναβαθμιστεί, να επεκταθεί αυτή η συνεργασία. Επίσης, πρέπει να δημιουργήσουμε και νέες μορφές συνεργασίας. Έχουμε εδώ το χέρι μιας γυναίκας. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερη ισορροπία μεταξύ των φύλων, χρειαζόμαστε περισσότερες γυναίκες στην ασφάλεια στον χώρο. και να χρησιμοποιήσουμε και τις νέες τεχνολογίες, την εκμάθηση μεσομηχανών για να βελτιώσουμε την αντίδρασή μας. Η έκθεσή μας αυτή για την αξιολόγηση απειλής είναι δημόσια, μπορείτε να την κατεβάσετε είναι περίπου 80 σελίδες ε, της έκθεσης. Αν σας ενδιαφέρει μπορείτε να τη διαβάσετε. Απαρτίζεται από διάφορα κεφάλαια και θέματα, οπότε σας ε, συστήνω την ανάγνωση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για την παρουσίασή σα και για τι εξηγήσει, κύριε Πρόεδρο. Και τώρα θα συζητήσουμε, όπω σα είπα, ο κύριος Στεχόφσκι θέλει να πάρει το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή. Ε, ενδιαφέρον παρακολουθείς αυτό που μας είπατε και κάθε χρόνο παρακολουθώ την ε, Παρουσίασε των ε, εκθέσεών σα. και πάντα προσβλέπω σε αυτές γιατί μας δίνουν μια καλύτερη εικόνα για το τι συμβαίνει πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Τρει ερωτήσει έχω να σα απευθύνω. Θα ήθελα να μου πείτε. Πώς λαμβάνει η χώρα αυτή η συνεργασία. οι ομάδες που διαθέτουν ε, προϊόντα παιδικής πορνογραφίας. Κάποιες ε, ΜΚΟ μας έχουν επισημάνει σε εκθέσεις τους ότι υπάρχει παιδική πορνογραφία από την Ασία, η οποία εισαγάγεται όλο και πιο πολύ προς την Ευρώπη. Και πραγματικά είναι τεράστια η αύξηση του όγκου της παιδικής προγραφίας. Τι γίνεται, για παράδειγμα, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τις ε, αστυνομικές αρχές της Κίνας. Ε, καταπολεμούνται αυτές οι πρακτικές οι οποίες προσωμιάζουν σε κυκλώματα μαφίας από πλευράς ε, συμμοριών της Κίνας ή άλλων συμμοριών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Δεύτερη ερώτηση. Τι ποσοστό επιτυχίας υπάρχει σε ό,τι αφορά τη σύλληψη εγκληματιών που χρησιμοποιούν ε, παραχαραγμένες ε, συνδέσμους, ε, διευθύνσεις IP και προβαίνουν σε παράνομες ενέργειες ό,τι αφορά τα κρυπτονομίσματα. Αναφέρατε συμμορίες από την Βεντική Αφρική, συνεργασία επίσης με την αστυνομία της Τσεχίας, γενικά η συνεργασία με τις αρχές των νέων κρατών μελών αποτελεί ένα θέμα. Τρίτο σημείο που ήθελα να ρωτήσω. Οι γενικές δραστηριότητες ε, από hackers της πρώην Σοβιτικής Ένωσης ε, στην Τσεχία. Είναι αυξανόμενη η δράση των Ρώσων hacker που προσπαθούν να εισβάλλουν ε, στις υποδομές και στα δεδομένα τσεχικών εταιριών. Παρακολουθείτε με επιτυχία τέτοιου είδους εγκλήματα. Ή δεν υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών σε αυτό το επίπεδο. Ευχαριστώ. Κύριε Δεχόφς ήταν αυτός. Κάνε μία άλλη ερώτηση. Θέλει να πάρει το λόγο. Κανεί άλλο. Αν όχι, να σα δώσω το λόγο για να απαντήσετε. Σα ευχαριστώ που μου δίνετε και πάλι το λόγο. Σα ευχαριστώ και για τι ερωτήσει σα. Για να δω τι σημειώσει μου. Η πρώτη ερώτηση σε ό,τι αφορά τη συνεργασία και πώ λαμβάνει η χώρα, πώ διαμορφώνεται αυτή η συνεργασία Νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια επιτυχία τη Europol και καλά θα κάνουμε το να, να το αναφέρουμε. Δεν ξεκινάμε δικέ μα έρευνε. υποστηρίζουμε όμω τα κράτη-μέλη και έχουμε μεγάλη επιτυχία στον τομέα αυτό. Αποτελούμε ένα κούμβο ε, μυστικών πληροφοριών και μια πλατφόρμα συνεργασία στην οποία όλοι οι φορείς μπορούν να συνεργαστούν. Όλοι λοιπόν μπορούν να υποστηρίξουν στα πλαίσια της εργασίας αυτής τις έρευνες και επιπροσθέτως... Α, έχουμε συστήσει συμβουλευτικές ομάδες με τον ακαδημαϊκό κόσμο, με τις ε, επιχειρηματικά συμβούλια, εταιρικά συμβούλια. Υπάρχει λοιπόν μια πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στο μοντέλο και διαφόρων άλλων μεγάλων εταιριών ε, στις κόλπους της Europol και έτσι λοιπόν όλες οι πληροφορίες, όλες οι μυστικές πληροφορίες που συλλέγουμε από τα κράτη-μέλη δεν είναι κατοχή, στην κατοχή μας, δεν είναι διεκτησία μας, αλλά συγκεντρώνεται στους κόμβους, στον κόμβο μας και έτσι νομίζουμε ότι το μοντέλο είναι επιτυχές για τη συνεργασία και για την ε, έκβαση των ερευνών. Το ίδιο συμβαίνει και στον τομέα της πρόληψης και της ευαισθητοποίησης. Έχουμε καλή συνεργασία και με τον εταιρικό κλάδο. Μία πρωτοβουλία θα ήθελα να αναφέρω την Νόρμα ε, Ράντσον με τι ε, Ολλανδικέ ε, Αστυνομικέ Αρχέ. Ξεκίνησε από την από 2-3 χρόνια με No More ονομάζεται λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία σε πολλές γλώσσες, σε πολλές πλατφόρμες, πολλές χώρες. Αποτελεί ένα πολύ καλό παράδειγμα του πώς συνεργούμε. Δεύτερο ερώτημα για την σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών online και το σχετικό πορνογραφικό υλικό. Βλέπουμε λοιπόν διάφορε τάσει στο σημείο αυτό. Όχι μόνο οι εγκληματίε που κάνουν κατάχρηση διάβλων επικοινωνία ε, για να διανέμουν τέτοιο υλικό, αλλά και του τόρ, αλλά και αυξανόμενη κατάχρηση. Ζωντανή εξαποστάσεως κακοποίηση παιδιών ε ζωντανή κακοποίηση παιδιών με βίντεο εφαρμογές, το οποίο αποτελεί μια πρόκληση. Θα καταλαβαίνετε όχι μόνο από τεχνικής άποψης πώς θα γίνει η σχετική έρευνα, αλλά πώς θα βρούμε και μεθόδου συνεργασία με τι χώρε στόχο. Εκεί που λαμβάνει η χώρα η εκμετάλλευση των παιδιών. Δεν είναι απλά τα πράγματα που καταλαβαίνετε, αλλά έχουμε διάφορε επιτυχίε και εδώ αναπτύσσουμε το δίκτυο συνεργασία μα. Αναφέρεται την Κίνα, Προφανώ. Δεν είναι άμεσα εταίρο μα η Κίνα. Έχουμε όμω κάνει επισκέψει και έχουμε και καλή συνεργασία. Και τουλάχιστον στον τομέα αυτό υπάρχει καλή συνεργασία σε επίπεδο εργασία. Η Ιντερπολ επίση αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο επίπεδο αυτό. Τι μπορεί να κάνει η Ιντερπολ για τα διδαχθεί αυτά εγκλήματα. Μια υποερώτηση, αν δεν κάνω λάθο, για το ποσοστό επιτυχία για τη σύλληψη εγκληματιών που χρησιμοποιούν ε, παραχαραγμένε ταυτότητε ε, και ε, χακάρουν πορτοφόλια και το καθεξή. Αυτό δύσκολα μπορώ να σα το απαντήσω σε ερώτημα. Γιατί όπω σα είπα, εμεί δεν Εκκινούμε δικέ μας έρευνες. Δραστηριοποιούμαστε μόνο σε έρευνες που συμπεριλαμβάνουν δύο και πλέον Ουσιαστικά θα έλεγα ότι βλέπουμε την κορυφή μόνο του παγόβουνου. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις, ναι, σημειώνουμε επιτυχίες. Αλλά γενικά αυτό αποτελεί μια πρόκληση για όλε τι αρχές επιβολής του νόμου. Η συνεργασία, όπως είπατε, αποτελεί πρόκληση κλειδί και αυτό ενδεχομένω να ενδιαφέρει και το ακροτήριό μας. Προσπαθούμε να καταρτήσουμε την τρίτη έκθεσή μας με την Europol σε ό,τι αφορά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην διεθνή συνεργασία. Τρίτο ερώτημα για τους hacker. Αυτό δεν είναι στο πεδίο εφαρμογής μας. Εμείς εστιαζόμαστε στην καταπολέμηση εγκλήματος, για τα κυβερνοεγκλήματα συγκεκριμένα. Αυτό θα πρέπει να το μεταφέρουμε ως ερώτημα στη πόλα. Αυτό εμπίπτει καθαρά στην εθνική αρμόδιότητα των κρατών μελών. Και σε καμία περίπτωση στο πεδίο εφαρμογή το δικό μας. Ερώτηση εκτός μικροφώνου. Δεν γνωρίζω. Απαντάει ο κύριος Αμάν. Ευχαριστούμε για τις εξήγησεις σας. Άλλες ερωτήσεις. Θέλει κανένα άλλος να πάρει το λόγο, να σχολιάσει. Αν όχι, να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, αν συμφωνείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αμάν. Το δεύτερο σημείο λοιπόν σήμερα το απόγευμα αφορά την εργασία της ομάδας εργασίας της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για τον έλεγχο στα πλαίσια του Σέγγεν. Παρουσίαση λοιπόν της ομάδας Βίσκος, ο κ. Καλός θα μας παρουσιάσει. Από την ομάδα για τον έλεγχο του Σέγγεν, για τον κρίσιμο ρόλο ευαισθητοποίηση για θέματα που αφορούν το Σέγγεν. Και η Επιτροπή μας έχει αρμοδιότητες ελέγχου. Ο κ. Σκοέλιο θα μας αναφέρει, θα μας παρουσιάσει την ε, παρέμβασή του και μετά το λόγο δικό σας. I am glad. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά σας αναφέρω ότι έγινε στην ομάδα εργασία για τον έλεγχο ε, Σέγγεν και πρόκειται για αυτήν την task force που συνεδρίασε κάθε μήνα και ενημερωνόμαστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσία του Συμβουλίου και των κρατών μελών και είχαμε και τους ε, διευθυντές της Europol, της Ακτοφυλακής και της Υπηρεσίας των Δικαιωμάτων. Επίσης, εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο η πρωτητήσια έκδοση για το, έκθεση για το Σέγγεν με πρωτοβουλία της ομάδας εργασίας και ήμουν συγκητής. Είχαν ρόλο κλειδί τα μέλη και η γραμματεία. Πολύ αποδοτική η ομάδα και μπράβο της. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σας πω ποια σημεία θεωρήσαμε πιο σημαντικά και εστιάσαμε την προσοχή μας. Πρώτα-πρώτα, όπως γνωρίζετε, η ομάδα εργασία συγκροτήθηκε για να εξασφαλίσει το πώς θα μπορέσουμε να ασκήσουμε το δημοκρατικό μας δικαίωμα του ελέγχου. Επίσης, τουλάχιστον σε μία περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας έδωσε πρόσβαση όπως και δώσει στα κράτη-μέλη το σου και η συμμελήψή του στα της ε, ακτοφυλακής ήταν η απόδειξη ότι ακόμα είμαστε απ' έξω. Και έτσι για το μέλλον του Eurosur στη σύντηση δεν είμαστε παρόντες και μόνο εκ των υστέρων το ανακαλύψαμε και επιμείναμε ότι θα πρέπει να συμμετάσχουμε τότε μόνο σε εκείνες τις συνεδριάσεις μας κάλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μεγάλο αυτό το επίτευγμα, αλλά φάνηκε ότι ακόμα πολλά πρέπει να γίνουν για να εξασφαλίσουμε ότι η Κομισιόν και το Συμβούλιο συμμορφώνονται με την υποχρέωση της ε, πίστης συνεργασίας και ότι δέχονται το Κοινοβούλιο ως αυθεντικό συνομοθέτη σε όλες τις φάσεις λήψης αποφάσεων. Κατά δεύτερο λόγο δεν θα σας εκπλήξω αν σας πω ότι οι έλεγχοι εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων παραμένουν ε, που σημείο το οποίο μας ενδιαφέρει και η αίτηση, γιατί η αιτήση έκθεση για το Σέγγεν ήταν ξεκάθαρη για τη θέση μας. Η σημερινή έλεγχη είναι παράνομη και παράλληλα κάποια κράτη-μέλη και δεν, και δεν αναφέρομαι στα κράτη-μέλη των εξωτερικών σύνορων δεν ε, τηρούν τις υποχρεώσεις τους για τα εξωτερικά σύνορα δηλαδή το να ελέγχονται όλοι. Και όπως λέει η έκθεση, το πρόβλημα παραμένει παρά τις προσπαθίες μας. Μην κάνουν τίποτα τα κράτη-μέλη και το αναφέραμε ότι το κοινοβούλιο δεν μπορεί άπρακτο να παρακολουθεί και να έχουμε αυτούς τους ιστορικούς ελέγχους. Κατά τρίτο λόγο, Καλέσαμε τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και μας ενημέρωσαν για το έργο τους, ανέγυψαν κάποια ζητήματα και τώρα πρόκειται να απευθύνουμε στον Επίτροπο Αβραμόπουλο μια επιστολή ζητώντας πρόσβαση στην ετήσια ανάλυση για το έγκλημα και για πιθανές παραδιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλες τέτοιες εκθέσεις της Επιτροπής και όχι του Κοινοβουλίου. Τέλος, μάθουμε ποια είναι τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ούτως ώστε να εξαιρέσει κάποιες υπηρεσίες από κάποιες εξελίξεις, κάποια διαβήματα. Τελευταίο θα πρέπει να καλύψουμε το Brexit και την μέλουσα σχέση όσον αφορά την ασφάλεια με την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν προκειμένου η Επιτροπή, αφού εμείς επιμείναμε, ενημέρωσε την ομάδα εργασία για την προσωρινή ε, άδεια χρησιμοποίηση του συστήματος ΣΑΙΑΣ από το Ηνωμένο Βασίλειο και έγινε σχετική συνάντηση παρουσία μας, γιατί όπως γνωρίζετε δεν είναι στο ΣΕΝΚΙ το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά έχει προσωρινή πρόσβαση στο σύστημα SIS, το σύστημα πληροφοριών, αστυνομική συνεργασία και όχι για τα εξωτερικά σύνορα, τα έλεγχο των σύνορων τέλο πάντων. Οπότε θα πρέπει να δούμε κατά πόσον τηρούν τα όσα προβλέπονται και τώρα ε, πρόκειται να υπάρξουν νέες συστάσεις. Ακόμη πάρα πολλά πρέπει να διευκρινιστούν, πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε κάνει το Συμβούλιο. Επιτρέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο να έχει πρόσβαση. Μα θα πρέπει τότε να συμμορφωθεί με τις συστάσεις του Ηνωμένο Βασίλειο. Τι να περιμένουμε ότι στο μέλλον εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βρίσκονται και ενώ τώρα δεν συμμορφώνονται αυτούς τους κανόνες που είναι μέλη της Ένωσης, δεν συμμορφώνονται τότε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα παρά ποτέ απειλείται το Σέγγεν. Άρα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτω ώστε να προστατεύσουμε την ακυρότητα της περιοχής του Σέγγεν ε, χώρου ελευθερίας και ασφαλείας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βλέπω ότι κάποιοι συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο, τουλάχιστον δύο από την Ομίγυρη, που ήδη ζήτησαν το λόγο. Άλλος κανείς παρακαλώ. Κύριε Γκόμες, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι και εγώ μέλος αυτής της ομάδας εργασίας, της οποίας προεδρεύει με ιδιαίτερη επιδεξιότητα ο Κάρλος Κοέλιο. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το έργο αυτής της ομάδας εργασίας και η συνεργασία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συμμερίζομαι πλήρως τα σχόλια του Προέδρου μας ομάδα εργασίας και επίση ασθενίζομαι τι ανησυχίε του σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και τις συνέπειες που θα έχει το Brexit ε, για τη, τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Αρχίζω και αποκαλύπτω πράγματα που με συγκλονίζουν και με ε, καταπλήσουν. Θα σταθώ σε τρία από αυτά. Ε, μία βασική χώρα, χώρα μέλος, δεν θα πω το όνομα, που λόγω του, της μελέτης ε, κινδύνου που έγινε από τις αρμόδιες αρχές αποφάσισε να μην χορηγήσει θεωρήσεις Σέγγεν σε κάποιους ε, πολίτες και παρόλα αυτά εξακολουθούν να βρίσκονται στην επικράτειά του και μέσω άλλων διάβλων, δεν ξέρω ποιον, καταφέρνουν να έχουν πρόσβαση στο χώρο Σέγγεν. Αυτό είναι πολύ σοβαρή, με τι άλλο, επικάλυψη των διάβλων. Κάτι που θα μπορούσε ίσως να υπονομεύσει και το ίδιο το σύστημα Σέγγεν. Δεύτερο ζήτημα μία υπόθεση που αφορά τη Μάλτα. Εδώ θα κατονομάσω τη χώρα. Και μάλιστα την επισήμανα όχι μόνο στην ομάδα εργασία ε, και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ένα σύστημα ε, που πουλά θεωρήσεις ε, Σέγγεν της Μάλτας για εξαγωγή χρημάτων. Και μάλιστα αυτές στείνονται σε πολίτες από τη Λιβύη, Αλγερία και μάλιστα μπλέκεται και το γραφείο του Πρωθυπουργού και οποιοδήποτε με θεώρηση από τη Μάλτα μπορεί να πάρει ένα ferry boat και σε λίγο καιρό να βρεθεί στην υπηρετική Ευρώπη, στην Ιταλία. Έχουμε καθημερινές συνδέσεις ε, με τη Μάλτα και μπορούν είτε με εθνική θεώρηση είτε με θεώρηση Σέγγε να μπουν στην υπηρετική Ευρώπη και ε, έγινε με δωροδοκία του Νάβελ Γκάφ ενός ε, αξιωματούχου γνωστού. Μάλιστα ήταν ειδικό απεσταλμένος τη κυβέρνηση τη Μάλτα, κάτι που το αρνήθηκε. Αλλά έτσι παρουσιάστηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωση τη Λιβύη και ο τρόπο που τον υποδέχτηκαν α, στη Λιβύη από τον Υπουργό Εσωτερικών και κάποιον άλλον έδειχνε ότι ήταν πραγματικά απεσταλμένος, ειδικός απεσταλμένος του Πρωθυπουργού της Μάλτας παρόλο που το διέψευσε το γραφείο του Πρωθυπουργού και παρά τα τεκμήρια και τα πιστήρια και τα στοιχεία που καταθέσαμε για το θέμα αυτό, και μάλιστα υπάρχει και σχετική δίκη που έχει ξεκινήσει στη Μάλτα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τα σχήρα τη, λέει ότι δεν γνωρίζει τίποτα και δεν ε, έχει δυνατότητα να το ελέγξει. Νομίζω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεχνά τι τεράστιο κίνδυνο δημιουργεί μια τέτοια κατάσταση. Είναι απαράδεκτη η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχω στα χέρια μου τη γραπτή απάντηση του Επιτρόπου Αβραμόπουλου. και το ακούσαμε και στην ομάδα εργασία από εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν δέχομαι αυτέ τι εξηγήσει που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν δέχομαι ε, αυτή την απόπειρα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανοίξει τα σχέδια και να αποποιηθεί των ευθυνών τη ε, σε ένα ζήτημα που διακυβεύει την ίδια την ακαιρεότητα του Σέγγεν, του συστήματο Σέγγεν. Μια τέτοια στάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απαράδεκτη. Και τρίτο θέμα, αφορά τη Σέουτα και τη Μελίγια. Έχουμε πάει και μαζί μάλιστα στη Μελίγια, όχι ακόμη στη Θέουτα. Και εκεί είναι πολύ προβληματική η κατάσταση, γιατί είναι τα μόνο δύο εδάφη, η Σέουτα και η Μελίγια, που βρίσκονται στη Βόρεια Αφρική και περιστοιχίζονται από τεράστιους φράχτες και με σειρματοπλέγματα ηλεκτροφόρα και παρόλα αυτά πολλά εγκληματικά κυκλώματα εξακολουθούν να διακινούν μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει ιδιαίτερα τις πανικές Αρχές που έχουν καταβάλει τεράστιες προσπάθειες και το έχουμε διαπιστώσει. Αλλά δεν έχουμε καμία ευρωπαϊκή αντίδραση από ευρωπαϊκά όργανα, τη Frontex για παράδειγμα ή ε, τη συνοριοφυλακή. Ενώ είναι ευρωπαϊκά τα σύνορα στη Θεότα και τη Μελίγια. Και με ενοχλεί αυτό και με ε, εκνευρίζει γιατί όλα όσα γίνονται στη Σεούτα και τη Μελίγια γίνονται επειδή είναι έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και, και λόγω του τρόπου που γίνονται οι έλεγχοι από τις εθνικές αρχές. Πάντω, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όπως η Frontex και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λάμπουν δια της απουσίας τους και αφήνουν τα πάντα στις εθνικές αρχές, στι Και στρέφουν αλλού το βλέμμα. Αυτό είναι πραγματικά εξοργιστικό. Για να μην μιλήσω για τις χρυσέ βίζε, για τις χρυσέ θεωρήσει. Και ακριβώς επειδή δεν έχουμε μητρό ε, που να καλύπτουν και τις ιδιωτικές πτήσεις. Το τι γίνεται και τι παραβιάζει του Σέγγεν λαμβάνουν χώρα στα κράτη-μέλη είναι τελείως εκτός ελέγχου. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα που χρήζει διαφορετική προσέγγιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γκόμες. Κυρία Ιντβελτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ σύντομα, γιατί συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με τα σχόλια της Άννας Γκόμες. Δηλαδή, η ακεραιότητα του χώρου Σέγγεν εξαρτάται από τη συμπεριφορά των κρατών μελών. Και αναφέρατε κανένα δύο παραδείγματα που είναι συζητήσιμη πολύ αυτή η συμπεριφορά. Για να μιλήσω για την Πολωνία, όπου το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν ε, είναι αντικείμενο κατάχρηση για την παρενόχληση μη κυβερνητικών οργανώσεων που επικρίνουν την κυβέρνηση. Οπότε εκεί χρειαζόμαστε ακόμη πιο ευρυθή συζήτηση. Την περασμένη εβδομάδα που σας παρουσιάσαμε την έκθεση αποστολή στην Μάλτα, ε, μίλησε για την ε, πώληση διαβατηρίων και αδειών ε, παραμονής που αμφιβάλλω αν συνάδων με το Σέγγεν. Ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και μια δυσκολία με τους ετούντες άσυλο για τους πρόσφυγες τους μετανάστες, αλλά τους στρώνουμε το κόκκινο χαλί και δεν ρωτάμε τίποτα ως μπορούν να εξαγοράσουν την είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ζήτησα από την ομάδα εργασίας να το εξετάσει. Επίσης, το Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίζει να έχει πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Είμαι κατά και θα πρέπει να επαγρυπνούμε. Θα συνεχίσουμε να είμαστε φίλοι και στενοί σύμμαχοι με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν μπορούμε να επιτρέψουμε και μετά το Brexit ε, ε, ανεξέλεγκτη εισαγωγή και χρήση των, ε, του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν. Ευχαριστώ. Κυρία Βερζά. Βερζιά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κάρλος Κοέλιο για το έργο του και την επιμονή του την αντοχή του και το διαλλακτικό του πνεύμα και την ικανότητα που έχει να φογκράζεται τους συναδέλφους. Συμφωνούμε, συμφωνούμε ως προς τους στόχους και αυτό μας διευκολύνει. Θα ήθελα να συγχαρώ και τη Γραμματεία για τη βοήθειά της και τη διευκόλυνση του έργου της ομάδας εργασίας. Νομίζω ότι Όλοι αγαπούμε το χώρο Σέγγεν και την ελευθερία διακίνησης που εξασφαλίζει. Αλλά αυτό που με τρομάζει, ε, ακόμη και μετά τη συμμετοχή μου στην ε, ε, ομάδα αυτής της εργασίας, είναι η, η χειραγώγηση, η κατάχρηση του συστήματος που κάνουν τα κράτη-μέλη, ο τρόπος το οποίο εργαλειοποιούν το σύστημα τα κράτη-μέλη και οι αδυναμίες που έχουν στη διαχείριση του συστήματος. Ελπίζω να βελτιωθεί αυτή η διαχείριση. Πάντως ε, αυτό που κατάλαβα είναι η ανεπάρκεια των μέσων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διενέργεια ουσιαστικών ελέγχων. Γιατί μας είπαν ότι ε, η έλεγχη αυτή ποτέ δεν είναι ευνίδη. απροειδοποίητη. Αν θέλουμε όμως πραγματικό και αποτελεσματικό έλεγχο, θα πρέπει να γίνονται ευνίδη έλεγχοι απροειδοποίητα και μάλιστα ανα πάσα στιγμή από ad hoc υπηρεσίες που θα έχουν τα κατάλληλα μέσα και τα εφόδια για να του πραγματοποιήσουν. Κάτι που δεν ισχύει δυστυχώ σήμερα. Ε, το δεύτερο δίδαγμα που άντλησα από τη συμμετοχή μου στην ομάδα εργασία είναι η διατήρηση των εσωτερικών ελέγχων. Και μάλιστα γίνεται μερικές φορές κακή διαχείριση αυτών των εσωτερικών ελέγχων από κάποια κράτη-μέλη, γιατί κάνουν του ελέγχους ε, για άσχετου λόγου. που παραβαίνουν αυτό το λόγο θέσπιση και επαναφορά των εσωτερικών ελέγχων. Δεν θα κατονομάσω συγκεκριμένες χώρες, αλλά ξέρουμε ότι γίνεται κατάχρηση αυτών των εσωτερικών ελέγχων και για λόγους που είναι άσχετοι με αυτούς για τους οποίους θεσπίστηκαν. Και μάλιστα με τρόπο που είναι επιζήμιος για το σύνολο του χώρου Σέγγεν και για την αξιοπιστία του χώρου Σέγγεν, κυρίως για τους πληθυσμούς των ε, ενδιαφερόμενων περιοχών. Σε ό,τι αφορά το Brexit και τα προβλήματα της Μεγάλης Βρετανίας, αυτό που έμαθα εγώ στην ομάδα εργασίας είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούσε πώς θα το πω, μονομερός το σύστημα πληροφοριών σε κάτι που δημιουργούσε ήδη πρόβλημα. Και το Συμβούλιο δεν ε, είχε μία ad hoc συμπεριφορά σε σχέση με το Brexit και την πίεση που θα προκαλούσε για το θέμα του συστήματος πληροφοριών Σέγγεν, θα συνεχίσουμε φυσικά να έχουμε χρήσιμες, ωφέλιμες σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, υπό τον όρο όμως ε, να, είναι, να δράζονται σε υγιείς βάσεις αυτές οι σχέσεις. Προς το παρόν δεν είναι υγιείς αυτές οι βάσεις συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Και θα ήθελα να επαναλάβω του φόβου μου για τη Βουλγαρία. Γιατί η Βουλγαρία είναι εκτό του χώρου Σέγγεν, αλλά πληρεί όλε τι προποθέσει για να ενταχθεί στο χώρο Σέγγεν αυτό που συμβαίνει στα σύνορα Τουρκίας και Βουλγαρίας ε, με προβληματίζει πολύ. Και μάλιστα συμμετείχα σε μια αποστολή στα σύνορα, στα βούλγαρο-τουρκικά σύνορα και ε, τα στοιχεία που λαμβάνουμε για όσους προσπαθούν να περάσουν αυτά τα σύνορα με κάνουν να αμφιβάλλω για τις δυνατότητες εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου, κυρίως ό,τι αφορά τους Τούρκους υπηκόους, που στα πλαίσια της ε, αποτελεσματικής αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας ίσως ζητήσουν άσυλο. Και τέτοια βουλγαροτουρκική αστυνομική συνεργασία ισχύει εδώ και 45 χρόνια. Τώρα όμως έχουμε κάποιες αλλαγές στο καθεστώς και δεν αποκλείεται να, ζητηθούν, ε, να ζητηθεί άσυλο από πολλούς Τούρκους υπηκόους θα πρέπει να φροντίσουμε να μην συρρυκνωθεί αυτό το δικαίωμα και να διαλευκάνουμε την κατάσταση στα τουρκοβουλγαρικά σύνορα. Επίσης, πιστεύω ότι θα ήταν κρίμα να μην έχουμε και γραπτή έκθεση, ένα έγγραφο εργασίας, ένα είδος απολογισμού του έργου αυτής της ομάδας εργασίας, για να μείνει κάποια παρακαταθήκη αυτή αυτής της προσπάθειας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί και στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία. Και ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή μας, τον κύριο Κουέλα. Σα ευχαριστώ για τα σχόλια σα, λέει ο Πρόεδρο. Και αν ε, δεν θέλει κανεί άλλο στο λόγο, μήπω να πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μα μιλήσει. Θα θέλετε να πάρετε το λόγο, να σχολιάσετε την ομάδα εργασία τη Επιτροπή μα σχετικά με τον έλεγχο του Σέγγεν. Ο κ. Ελιβιέ Σεπχαρτ είναι εδώ από τη Γενική Διεύθυνση Home. Θα θέλετε να πάρετε το λόγο. πρώτο δώσουμε πάλι το λόγο στον εισηγητή μα τον κύριο Κόλιο. Σας ευχαριστώ και καλησπέρα σας. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι χαρά μας να συνεργαζόμαστε με τον κύριο Κοέλιο και την ομάδα ελέγχου του. Νομίζω ότι οι συζητήσεις αυτές είναι αμοιβαίως υποφελείς και πραγματικά προσπαθούμε να διαβιβάσουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε σε ό,τι αφορά το Σέγγεν. Γνωρίζοντας ότι το Κοινοβούλιο και ο κύριος Κοέλιο είναι μεγάλοι προασπιστές του χώρου Σέγγεν, συχνά τον τελευταίο, τα τελευταία χρόνια έχουμε ακούσει ότι ο χώρος Σέγγεν είναι υποκίνδυνο. Είπατε, αναφέρατε την ομάδα εμπειρογνωμόνων, κύριο Σούρτ, εγώ το 2011-2012 συμμετείχα σε αυτήν την ομάδα όταν προετοιμάσαμε το Eurosur και τη σχετική νομοθεσία. Τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Γραμματεία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ προσκλήθηκε και συμμετείχε στην ομάδα αυτή τακτικά. Τι έγινε το 2017 όταν πάλι διοργανώθηκε η ομάδα αυτή με εκπροσώπους των κρατών μελών. Από πλευράς μας επιμείναμε σε κάποια χρονική στιγμή να ακολουθηθεί η διαδικασία. Απλά χρειαζόταν μια επίσημη, ένα επίσημο αίτημα από πλευρά του Κοινοβουλίου για να συμμετέχει στην ε, διαδικασία. Μόλι λάβαμε λοιπόν αυτό το επίσημο αίτημα από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του. Λυπάμαι αν υπήρξε παρανόηση. Αλλά αυτή ήταν η αλήθεια. Πάντα ήμασταν ανοιχτοί στη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ομάδα αυτή. Κλείνοντα, να πω ότι ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία και νομίζω ότι θα χρειάζεται ακόμα πιο πολύ στους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Ακόμα πιο πολύ από ό,τι στην αρχή, γιατί το Σέγγεν δυστυχώς εξακολουθεί να μην είναι πλήρες ακούμε ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε στο Σέγγεν. Είμαστε ακόμα στο Σέγγεν. Δεν έχουμε απομακρυνθεί από το Σέγγεν, αλλά θέλουμε να επανέλθουμε σε μια φυσιολογική λειτουργία του Σέγγεν. Ελπίζουμε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή. Και σα ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Σέφερτ. Ο κύριο Κοέλιο. Θέλετε να πάρετε το λόγο να κάνετε κάποια καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, να ευχαριστήσω τα μέλη της ομάδας εργασίας. Είναι πολύ καλή η ομάδα μας. Και προσπαθούμε να εκπληρώσουμε αυτά που μας έχει ζητήσει η Επιτροπή να κάνουμε. Κατά δεύτερον, να συνεργαστούμε για τα θέματα τα οποία έχουμε ακόμα επιτάπητος. γιατί ακόμα πρέπει να διευκρινιστούν κάποια εκκρεμή ζητήματα για να εξασφαλιστεί ο κοινοβουλευτικό μα έλεγχο. Και κατά τρίτον, θα ακολουθήσουμε την πρόταση τη κυρία Βερζιά. προκειμένου να καταγράψουμε σε χαρτί όλα μας τα πορίσματα για το επόμενο κοινοβούλιο κατά πάσα πιθανότητα το χρονοδιάγραμμα μας δεν θα μας επιτρέψει και άλλη μία έκθεση, μια και ζητήσαμε πέρσι έκθεση, αλλά νομίζω ότι τουλάχιστον τον τρόπο αυτό ε, εξασφαλίσαμε μία μέθοδο διαφύλαξης των εργασιών μας και για το επόμενο κοινοβουλίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας ευχαριστώ και για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε κύριε Κόλια. Σα ευχαριστούμε για την ηγεσία που επιδεικνύεται στον τομέα αυτό και δεδομένου του ότι το επόμενο ζήτημα είναι για τις 4.45 ε, και έχουμε ακόμα μισή ώρα, προτείνουμε ένα διάλειμμα, ένα σύντομο διάλειμμα μισή ώρας. Δεν βλέπω και την κυρία Μέτσολα εδώ. Το επόμενο θέμα είναι και πάλι για το Σέγγεν σε ό,τι αφορά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία και το σύστημα πιστοποίησης, ε, επαλήθευσης που χρησιμοποιείται στις χώρες αυτές. 16 και 45. Άρα θα έλεγα να κάνουμε ένα διαλυματάκι μισής ώρας. Θα Τα λέμε λοιπόν και 45.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 Υπότιτλοι the Well... Πρόεδρος, επιστρέφουμε στα καθήκοντά μας, στην συνεδρίασή μας και πάμε στην κοινή συζήτηση των σημείων υπαριθμών 5 και 6. Συνδυασμός των εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς Κοινοβούλιο και Συμβούλιο για Πρόοδο της Βουλγαρίας στο πλαίσιο μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου με την αντίστοιχη έκθεση για την πρόοδο της Ρουμανίας. Από την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των δύο χωρών τον Ιανουάριο του 2007 ε, θέσπισε αυτόν τον μηχανισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως έναν μηχανισμό για να βοηθήσει τις χώρες να διορθώσουν ε, κάποια κακώς κείμενα για τη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα για την περίπτωση της Βουλγαρίας για να αξιολογείται και επιτευχθήσα πρόοδος. Έχουμε εδώ για να μας ενημερώσουν ε, για τα όσα συζητήθηκαν στις 13 Νοεμβρίου τρέχοντος έτους τον διευθυντή από την Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Επιτροπής. Έχετε το λόγο. και στη συνέχεια θα υπάρξει συζήτηση για το θέμα μας. Και σας λέτε και το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και πάλι ευχαριστώ την Επιτροπή σας που δίνετε στην Κομισιόν την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε τις απόψεις μας. Πρώτα πρώτα να θυμηθούμε το πλαίσιο αυτών των εκθέσεων. Ξεκινούμε με την έκθεση του Ιανουαρίου του 2016 και Είπαμε ότι τώρα θα έχουμε μια γενική έποψη μιας δεκαετίας. Οπότε, κατόπιν τη αποφάσεις, άλλαξαμε την προσέγγισή μας. Πρώτα-πρώτα, είναι περιορισμένες οι συστάσεις που διατυπώνονται, αλλά είναι εφικτό να υλοποιηθούν πριν το τέλος της θητείας μας της Επιτροπής Επίσης, εστιαζόμαστε στο πώς μπορούμε να έχουμε κάποιες δομές, ούτως ώστε να στηριχθούν οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Εάν υπάρξει ε, πρόοδος, θα λάβουμε υπόψη τι μπορεί να γίνει για να μην έχουμε πίσω γύρισμα. Αυτά για αυτές τις δύο εκθέσεις. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πρόοδος σε σχέση με τις εστάσεις του Ιανουαρίου του 2017 και δεύτερον να δούμε κατά πόσον έχει υπάρξει κάποιο πίσω γύρισμα που έθεσε ένα αμφιβόλο την θετική αξιολόγηση του Ιανουαρίου του 2017. Όπως πάντα Κοστίζουμε πολύ προσεκτικά και τεκμηριωμένα και πρώτα πρώτα για την Βουλγαρία εν προκειμένου βλέπουμε σημαντικές προσπάθειες για υλοποίηση των συστάσεων και το συμπέρασμα είναι πως ενώ δεν τα έχουν καταφέρει 100% τα πράγματα βρίσκονται σωστή τροχιά και οι συστάσεις αφορούν τρία βασικά σημεία και θεωρούνται ότι σχεδόν έχουν υλοποιηθεί. Αυτά όσον αφορά την πρόοδο συστάσεις όπως το Ανώτοτο Δικαστικό Συμβούλιο, τις τροποποίησεις του ποινικού κώδικα και εμείς παρακολουθούμε την εξέλιξη για να μπορούμε να αξιολογήσουμε επίσης όσον αφορά τις συστάσεις ε, θα πρέπει να δούμε τι έγινε όσον αφορά την διαφθορά, τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και τη διαφθορά υψηλού επίπεδου. Οπότε είναι σημαντικό εδώ να καλύψουμε το θέμα του ότι η καινούργια υπηρεσία ε, κατά της διαφθοράς που αποτελεί μια καινοτομία τα τελευταία χρόνια ότι θα εδραιωθεί ως θεσμικό όργανο και θα συμβάλλει στον στόχο, δηλαδή να βελτιώσει τις επιδόσεις της ε, χώρας για την καταπολέμηση της εθρώσης ψηλού επίπεδου. Βέβαια δεν είναι μόνο αυτή η υπηρεσία, αλλά είναι βασικός της ρόλος. Επίσης, λέμε στην έκθεση ότι θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις ε, εξελίξεις και την πρόοδο και θεωρούμε ότι αν υπάρχει αυτή η θετική στάση, εάν ε, συνεχίζεται η εκπλήρωση των συστάσεων, η Βουλγαρία θα μπορέσει πριν το τέλος της ε, ε, θητείας μας να έχει ολοκληρώσει τα του μηχανισμού συνεργασίας και έλεγχου. Τώρα για τη Ρουμανία τα πράγματα είναι λίγο πιο περιπλεγμένα, είναι προκειμένου. Έχουμε το ζήτημα που διευνήσαμε το κατά πόσον υπάρχει πίσω κύρισμα όσον αφορά την θετική πορεία που είχε διαπιστωθεί ότι υπάρχει τον Ιανουάριο του 2017 και διαπιστώσαμε ότι έχει υπάρξει πρόοδο σε διάφορα μέτωπα. Το δε Νοέμβριο του 2017 στη σχετική έκθεση είχαμε επισημάνει τον κίνδυνο ότι ξανανοίγουν κάποια μέτωπα που είχαν κλείσει τον Ιανουάριο του 2017. Οπότε, κατά κάποιο τρόπο, αυτό προδίκασε το προηγούμενο της σημερινής έκθεσης και δεν έχει περάσει, δεν έχει αρθεί το σημερινό μας εκείνο και έχουμε συστάσεις για τρία μέτωπα πρώτα-πρώτα για την νομοθεσία όσον τη δικαιοσύνη για τον διορισμό των δικαστών και για τον ποινικό κώδικα ή τους κώδικες. Θέλουμε να επανέλθει στη σωστή πορεία η χώρα. Θα πρέπει να ξαναεξετάσουμε τα σχετικά μέτρα. Να δούμε τι γίνεται με τις συστάσεις. Να λάβουμε υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Βενετίας Επίση το Συμβούλιο, την ομάδα Γκρέκο τέλο πάντων που είναι κάποια ομάδα κρατών για την διαφθορά και συνενετικά είπαμε ότι θα πρέπει να ξαναλάβει την θέση που είχε θεσμικά το Ανάτοτο Δικαστικό Συμβούλιο. στην έκθεση. Μπορεί να δείτε ότι ξαναγίνεται κάποια ανάλυση των συστάσεων του νερού του 17. Μία-μία και της ε, επισυναπτωμένης τεχνικής εκθέσεως. Και έχουμε κάποια θεσμικά όργανα που ακόμα δεν έχουν παγιωθεί όπως για κάποια περιουσιακά στοιχεία. Ε, εκεί δεν έχει γίνει πρόοδος όσον αφορά τις 12 συστάσεις. Πρέπει να τονίσουμε ότι τα συμπεράσματα της Επιτροπής αποτελούν σημείο συμφωνίας όλων των παρατηρητών. Έχουμε προβεί σε δημοσιοποίηση δύο γνωμοδοτήσεων, πρώτα-πρώτα για την ταράθμιση της δικαιοσύνης και οι άλλοι για τους ποινικού κώδικες. Αυτά βοήθησαν Και όλα αυτά συνάδουν προς ε, το έργο της Επιτροπής της Βενετίας. Και επίσης ε, έχει ληφθεί υπόψη και η έκθεση του Κοινοβουλίου των Αρχών Νοεμβρίου. Βεβαίω και είμαστε ανοιχτοί σε περαιτέρω διάλογο και συνεργασία όσον αφορά τις ε, συστάσεις, αλλά θα πρέπει η Ρουμανία να επανέλθει στη σωστή τροχιά όσον αφορά την καταπολέμηση της διαφθοράς και όσον αφορά την ε, δικαστική μεταρρύθμιση. Επίσης, για τα επόμενα βήματα και σε σχέση με τις μέλουσες εκθέσεις είπαμε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διετίας θα προβούμε και σε νέα αξιολόγηση. Και σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Σλέης, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Με βάση το άρθρο 206 ε, επιτρέπεται και σε μέλη άλλων επιτροπών και όχι μόνο στα μέλη της ΛΥΜΠΕ να λάβουν μέρος στη συζήτηση ζητώντας το λόγο. Ο Πάβελ ζήτησε πρώτο το λόγο. Εδώ είμαι. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους συναδέλφους. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε. Αλλά περιμένω συγκεκριμένες απαντήσεις, όχι γενικές και αόριστες απαντήσεις σε ερωτήσεις, τότε θα είναι πραγματικές ευχαριστίες. Ξεκινώντας από το 2010, η Ρουμανία δεν έχει εμ, νομικές υποχρεώσεις ό,τι αφορά το CVM. Οπότε, τι άρθρο ε, στη συνθήκη υπάρχει για το CVM, για το Μηχανισμό Συνεργασίας και Ελέγχου. Ποια είναι η νομική βάση. Στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεπερνάει κατά τη γνώμη μου τις αρμοδιότητες που της εκχωρεί η συνθήκη. Δεν μπορείτε να θεσπίσετε τέτοιο μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου CVM μόνο για δύο κράτη-μέλη. Αν σας αρέσει τόσο πολύ ο μηχανισμός, τότε γιατί δεν τον εφαρμόζετε σε όλες τις χωρες μελη και στι 28 και εντό ολίγου 27. Και να ζητάτε από τη Ρουμανία να μην εφαρμόζει νόμους που έχει ψηφίσει η Βουλή και εγκρίνει το συνταγματικό δικαστήριο και κυρώσει το συνταγματικό δικαστήριο είναι παρέμβαση στα εσωτερικά μιας χώρας και υπαγόρευση σε μια χώρα τι να κάνει. Είναι απαράδεκτη αυτή η εμπλοκή σας στα εσωτερικά της Ρουμανίας. Επίσης αναφέρεστε συγκεκριμένους ανθρώπους. Μιλώ για το διορισμό του αρχισαγγελέα τη Εθνική Διάθεση κατά πολέμηση διαφθορά. και ζητείτε, ζητάτε αναστολή της διαδικασίας. Παρόλο που δεν έχει γνωμοτήσει ακόμη ο πρόεδρος, ζητάτε αναστολή της διαδικασίας απόλυσης του αρχισαγγελέα. Παρόλο που έγινε πολύ νομότυπα αυτή η απόλυση βάσει της αρμοδιότητας του Υπουργείου και του Υπουργού Δικαιοσύνης προωθείτε κάποιον και απαξιώνετε κάποιον άλλον. Είναι απαράδεκτη αυτή η ανάμειξή σας στα εσωτερικά της Ρουμανίας. Στη Γερμανία, μετά από μία μέρα απολύθηκε ο Γενικός εισαγγελέα. επειδή επέκρινε τον Υπουργό Δικαιοσύνη της Γερμανίας. Εκεί γιατί δεν είπατε τίποτα. Γιατί εφαρμόζετε διπλά μέτρα και σταθμά στι χώρε μέλη. Θέλω συγκεκριμένε απαντήσει. Επικρίνατε και άλλα νομοσχέδια που όμω εγκρίθηκαν από τη Βουλή τη Ρουμανία και εγκρίθηκαν και συνταγματικά από το Συνταγματικό Δικαστήριο. Πώ είναι δυνατόν να τολμάτε να ζητάτε από τη Ρουμανία να μην εφαρμόσει αυτού του νόμου ή να δίνετε εντολέ στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο της Ρουμανίας που έχετε επενέσει στο παρελθόν. Ζητάτε από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να αλλάξει τον επικεφαλής της δικαστικής επιθεώρησης και μάλιστα μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, ε, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο έστειλε επιστολή στην οποία αναφέρει ότι ζητήθηκε η θέσπιση της δικαστικής επιθεώρησης για να δοθούν εχέγγυα για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και των δικαστών. Αυτή ήταν η απάντηση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου μετά τη δημοσίευση της έκθεσής σας που δείχνει ότι ψεύδεστε. Ο μηχανισμός ε, συνεργασίας και ελέγχου αναφέρει την τη σύσταση αναστολής ε, κάποιων νόμων λόγω του, των ενεργειών του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, που είναι ο εγγυητής της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας, είχε μια θετική στάση και υπέβαλε προτάσεις για να βελτιωθούν οι νομικές διατάξεις. Και μάλιστα μερικές τέτοιες νομικές διατάξεις εγκρίθηκαν. Και εσείς το αμφισβητείτε αν διαψεύδοντας τον Νότο Δικαστικό Συμβούλιο που λέει ότι έγιναν δεκτές πολλές προτάσεις του και οι συστάσεις του περιλήφθηκαν στην Εθνική Νομοθεσία. Ποιος σας τροφοδοτεί με τέτοιες ψευδείς πληροφορίες που αποτελούν τη βάση για τις εκθέσεις σας. Γιατί έχετε μεροληπτικές πηγές για τις εκθέσεις σας και γιατί δεν ακούτε τα θεσμικά όργανα που υποτίθεται ότι κόπτεστε να ενισχύσετε. Πείτε μας ποιες είναι οι πηγές σας, πώς στοιχειοθετείτε τις εκθέσεις σας, πώς τις τεκμηριώνετε. Και επαναλαμβάνω, είναι απαράδεκτο αυτός ο πολιτικός μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου να εφαρμόζεται μόνο για δύο χώρες μέλη. Και αποσυστικά είναι αντικείμενο πολιτική χειραγώγηση από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη που δεν θέλουν τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία στο χώρο του Σέγγεν, φοβόμενοι ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα. Επίσης, ε, κάποιοι ηγέτες ε, χωρών που δεν θέλουν τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία στο χώρο Σέγγεν ακριβώς αυτό λένε. Στο μέτρο που ισχύει ο μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου, ξεχάστε την είσοδο στο χώρο Σέγγεν στη Βουλγαρία και Ρουμανία. Και εσείς λέτε δεν ισχύει κάτι τέτοιο, δεν σας πιστεύω όμως. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που ρωτήσατε τη Ρουμανία. Ζητήσατε από τη Ρουμανία να μην εφαρμόζει ε, τις αποφάσεις του Κοινοβουλίου της και την ομολογία του συνταγματικού της δικαστηρίου και να αναστείλει την απόλυση του Προέδρου της Εθνικής Διεύθυνσης Καταπολέμησης Διαφθοράς. Πώς είναι δυνατόν έτσι να ισχύει το κράτος δικαίου. Όλα, όλη αυτή η συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τροφοδοτεί αντιευρωπαϊκές τάσεις στη Ρουμανία γιατί τώρα ο κόσμος βλέπει πως χρησιμοποιούνται με πολιτικά κίνητρα αυτοί οι μηχανισμοί, φυσικά και ο κόσμος θα αντιδράσει και θα στραφεί κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε ίση μεταχείριση, ισότιμη με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Έχουμε τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις, αλλά όχι περισσότερα, περισσότερες. Συγγνώμη, παρακαλώ να είστε μετρημένοι στην τήρηση του χρόνου για να μην έχουμε υπέρβαση του ωραρίου της συνεδρίασης. Παρακαλώ, συνάδελφος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο, η έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντικατοπτρίζει την επιθυμία όλων των θεσμικών οργάνων της ε, Βουλγαρίας για την μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης και βλέπουμε ότι τρεις από τους έξι δείκτες θεωρούμε ότι έχουν ήδη κλείσει. Πρόκειται για τα έξι κριτήρια αναφοράς που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Τρία τέτοια κριτήρια έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Οπότε θεωρητικά η Βουλγαρία μπορεί να διεκπαιρεώσει το μηχανισμό συνεργασίας και ελέγχου στη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης είπα ότι είναι μία αναστρέψιμος αυτός, είναι μία αναστρέψιμη αυτή η πορεία. Επίσης και η συμμετοχή της Αγγελίας ήταν πολύ θετική και αναγνωρίζεται αυτό από την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βλέπουμε ότι έχουν δοθεί τα εχέγγυα για τη διαφάνεια του Γραφείου του Εισαγγελέα. Σε ό,τι αφορά το οργανωμένο έγκλημα, Έγιναν πολλές έρευνες εις βάρος ε, ε, υψηλά είσταμένων των βουλγαρικών αρχών κάτι που δείχνει πόσο καλά λειτουργεί το δικαστικό σύστημα στη Βουλγαρία και άρα ο μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου μπορεί να τερματιστεί του χρόνου. Και από τη στιγμή που θα εκπνεύσει αυτός ο μηχανισμός για τη Βουλγαρία, ελπίζω να μην χρησιμοποιήσετε προσχήματα για να αρνείστε ακόμη τη συμμετοχή της Βουλγαρίας στο χώρο του Σέγγεν. Ο κύριος Ράντεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντικειμενική της έκθεση. Οι συστάσεις της έκθεσης ε, από τον Ιανουάριο του 2017 έστειλαν το σαφές μήνυμα ότι μετά την ε, εφαρμογή των συστάσεων ο μηχανισμός συνεργασίας και ελέγχου θα έρθει σε αίσιο πέρας. Και μάλιστα ε, τον Νοέμβριο του 2017 αναγνωρίστηκε με, σε έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι πληρούνται τα κριτήρια ε, του 2017 και άρα δεν χρειάζεται να προσταθούν νέα κριτήρια. Και μάλιστα στην έκθεση του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με ε, τα κριτήρια αναφοράς του 2017 και τρεις από τους έξι δείκτες έχουν κλείσει προσωρινά, έχουν εφαρμοστεί. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι αν η Βουλγαρία συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό την πρόοδο και τι μεταρρυθμίσει, ο μηχανισμό συνεργασία και ελέγχου για τη Βουλγαρία θα έρθει σε πέρας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρόλο που υπάρχει θετική στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν είναι σίγουρο ότι τα κράτη-μέλη θα συμφωνήσουν με την εκπνοή του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου παρά την πλήρωση των κριτήριων από τη Βουλγαρία. Γιατί εξακολουθούμε να ακούμε τις εκκλήσεις πολλών κρατών μελών ε, να συνεχιστεί η εφαρμογή του μηχανισμού συνεργασία και ελέγχου χωρί καταληκτική προθεσμία. Και αυτό μπορεί να δικαιολογούνταν πριν από 10 χρόνια, αλλά όχι πια. Επίση, γίνεται κοινή συζήτηση Ρουμανία και Βουλγαρία, κάτι που είναι απαράδεκτο, γιατί είναι πολύ διαφορετική η πρόοδο των δύο χωρών και το περιεχόμενο των αντίστοιχων εκθέσεων. Άλλωστε, ο μηχανισμό συνεργασία και ελέγχου, όπω σχεδιάστηκε, δεν οδήγησε απτά αποτελέσματα. Χρησιμοποιήθηκε για πολύ καιρό ω πρόσχημα για πολιτικές επιθέσεις και βάση για πολιτικές επιθέσεις βάρος των δύο χωρών, παρά την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Η πατρίδα μου θα συνεχίσει να εφαρμόσει τι συστάσει και τι απαραίτητε μεταρρυθμίσει. Θα πρέπει όμω τα επιτεύγματα αυτά να αναγνωριστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τεθεί σε ένα τέρμα ο μηχανισμό συνεργασία και ελέγχου μετά την εφαρμογή και των τριών τελευταίων συστάσεων. Οτιδήποτε άλλο θα συνιστά διπλά μέτρα και σταθμά ει βάρο τη Βουλγαρία από του υπόλοιπου εταίρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, θα καταστεί σαφές ότι κάποιες χώρες μέλη δεν θέλουν τη Βουλγαρία στο χώρο του Σέγγεν. Αν κρίνουμε από τον συζητήσιμο νομικό δεσμό μεταξύ του Μηχανισμού Συνεργασίας και Ελέγχου και της ε, εισόδου μας, της ένταξής μας στο χώρο του Σέγγεν. Ε, κάτι τέτοιο είναι μια κατάφορη διάκριση βάρους βάρος της Βουλγαρίας, κάτι απαράδεκτο φυσικά για μας. Σα ευχαριστώ. Σχόλια από του συναδέλφου. κανεί άλλο θέλει να πάρει το λόγο. Η κυρία Στίβεν θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Ολλανδικά θα μιλήσω. Από αυτά που μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταλαβαίνω ότι είναι η 12η φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέταξε έκθεση σε ό,τι αφορά στα πλαίσια του, οργανισμού, του Μηχανισμού Συνεργασία και Ελέγχου και ζητά λοιπόν στην έκθεση αυτή η καλύτερη, διαπιστώσε μάλλον καλύτερη κατάσταση και στην Βουλγαρία και στην Ρουμανία. Αυτό προφανώ και αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα. Η κατάσταση λοιπόν έχει βελτιωθεί σε ό,τι αφορά το κράτο δικαίου. Και αυτό πραγματικά ήταν ε, σημαντική εξέλιξη και το οφείλουμε αυτό και στις ε, εκθέσεις, προσβλέπουμε και στο μέλλον σημαντικές εξελίξεις. Σήμερα λοιπόν έλαβα και ένα email από την κυρία Φανκέρκεν, η οποία αναφέρει ότι ενδεχομένω να υφίσταται ζήτημα στη Βουλγαρία σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της άνεξη θρησκείας, την αναγνώριση των θρησκειών και ότι η ενδεχομένω να υπάρχει πρόβλημα και σε ό,τι αφορά την αναγνώριση τη ατλαντική ε, εργασία και ενδεχομένω να κλείνουν μικροί ναοί. Θα μπορούσατε να μα δώσετε λίγο επιπρόσθετε πληροφορίες από αυτό. Ευχαριστώ. Okay, a very specific question. Μάλιστα, πολύ συγκεκριμένο ερώτημα, λέει ο πρόεδρο. Άλλο σχόλιο. Αν όχι, να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ακούσατε τα μέλη της Επιτροπής μας σε ό,τι αφορά το μηχανισμό ελέγχου και σταροποίησης της Ρουμανίας. Θα θέλετε να πάρετε το λόγο για να απαντήσετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω. Χαίρομαι που μπορώ εκ νέου να σας εξηγήσω από πού προέρχεται ο μηχανισμός ελέγχου και ε, συνεργασίας. Ξεκίνησε λοιπόν όταν ε, συμφωνήθηκε, όταν συνάφθηκε και συμφωνία προσχώρησε Οι δύο αυτοί μηχανισμοί προσθέθηκαν στην συμφωνία ως δεκλίδα ασφαλείας, αν θέλετε. Μια δεκλίδα ασφαλείας και προφανώς ε, μετά από δύο χρόνια δεν μπορούσαν να ισχύσουν ακόμα αυτές οι δικλείδες ασφαλείας. Δεν θα μπορούσαν να εφαρμοστούν καινούριε δικλείδες ασφαλείας, αλλά θα μπορούσαν να συνεχίσουν να υφίστανται οι παλιέ ε, τέτοιε ε, δικλείδες. Ε, υπήρχε λοιπόν ήδη ο CVM και εξακολουθεί να εφαρμόζονται σε ό,τι αφορά και τις ε, δύο χώρες. Αυτό λοιπόν ε, δεν άλλαξε. Η προσέγγιση τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επίσης δεν ε, τροποποιήθηκε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να σκητά τα καθήκοντα τα οποία της ανατέθηκαν στα πλαίσια του μηχανισμού CVM τα τελευταία 12 χρόνια με τον ίδιο τρόπο, με πειθαρχία και μετά από επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς οι οργανώσεις όπως η Επιτροπή της Βενετίας και τα άλλα κράτη-μέλη συμφωνούν σε γενική γραμμή με την ανάλυση της ε, κατάστασης όπως παρουσιάζεται στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είναι πεπισμένη ότι τα πορίσματα που αναφέρει στην έκθεση είναι καλά τεκμηριωμένα. Σε ό,τι αφορά τώρα αυτό που έχω να πω είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν και είναι σαφέστατη εδώ και χρόνια. Σε ό,τι αφορά το προηγούμενο που θα μπορούσε να δημιουργηθεί, δεν αποδεχόμαστε την αιτιολόγηση και τη σύνδεση που κάνουν διάφορε ό,τι αφορά το μηχανισμό συνεργασία και ελέγχου. Δεν θεωρούμε ότι δικαιολογείται το γεγονό ότι κατηγορούμαστε για ύπαρξη τέτοιας, ε, τέτοιου συνηθικού κριτικού. Δεν δεχόμαστε από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύπαρξη τέτοια σύνδεση. Κατά πόσον τώρα ο μηχανισμός ε, έχει οδηγήσει σε οποιαδήποτε βελτίωση. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασφαλώς και θεωρεί ότι έχει οδηγήσει σε βελτίωση. Η πρόοδος η οποία έγινε και η οποία σημειώθηκε στις εκθέσεις ε, του Ιανουαρίου του 2017 αποτελεί τεκμήριο για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί δεν πρόκειται για πανάκια σε καμία περίπτωση. Ούτε υποστήριξε ποτέ κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πρέχει όλες τις απαντήσεις, ούτε άλλωστε παριστάνει ότι ο σκοπός είναι να είναι απόλυτα τέλεια τα κράτη-μέλη. Ο σκοπός των οποίων είχε πάντα στο μυαλό της Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να επιτευχθεί μια κατάσταση η οποία θα είναι συγκρίσιμη, εύλογα συγκρίσιμη, με αυτή που επικρατεί σε άλλα κρατημέλη. Και νομίζω ότι τον Ιανουάριο του 2017 στην έκθεσή μας ε, το καταστήσαμε εξίσου σαφές και αυτό. Επίσης, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι οι εκθέσεις ε, CBM έχουν να κάνουν με περιορισμένο αριθμό τομέων σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση τη διαφθορές ε, και τις σχετικές μεταρρυθμίσεις. Δεν πραγματεύονται όλα τα αντικείμενα. Και για παράδειγμα, η ερώτηση αναφορικά με τους ναούς, ένα θέμα προφανώς θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν γνωρίζω την ε, συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά προφανώς είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Δεν εμπίπτει ωστόσο στον τομέα αρμοδιοτήτων της έκθεσης. Αυτά τα στοιχεία είχα να σας αναφέρω και ελπίζω να σας βοήθησα στο έργο της Επιτροπής. Μάλιστα, λέει ο Θέλει κανεί να απαντήσει στα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Πάβελ. Πάρτε το λόγο, αλλά σύντομα παρακαλώ. Η... Όπως και τι προηγούμενε χρονιές, δεν ναι, μου απάντησαν με συγκεκριμένο τρόπο στι ερωτήσει που έκανα. Ακούσαμε μόνο μία ομιλία, μία λιγόλεπτη ομιλία, η οποία ουσιαστικά αποφεύγει την ουσία. Δεν γίνεται αναφορά στις ε, μυστικές συμφωνίες μεταξύ μυστικών υπηρεσιών και δικαστικού σώματος, ε, συμφωνίες ε, που ουσιαστικά υπάγουν τους εισαγγελείς και τους δικαστές στις μυστικές υπηρεσίες. Γιατί δεν γίνεται αναφορά στις συμφωνίες αυτές, γιατί δεν τις καταδικάζουμε, γιατί αυτές οι συμφωνίες νικηβεύουν την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος στη Ρουμανία. Θα ήθελα να απαντήσετε παρακαλώ τις ερωτήσεις μου, όπως και τις άλλες ερωτήσεις που σας έκανα. Ο κύριος Λέιτ ήταν ξεκάθαρο σε ό,τι αφορά τις ε, απαντήσεις τους. Αν έχετε κάποια απάντηση όμως την εκτιμούσαμε. Πολύ ευχαρίστως. Απλώς τι απάντηση. Απλώ θα ήθελα να πω στον κύριο Παύλα, να κοιτάξει τη σελίδα 2 της έκθεσης. Έχω μια εκτενή παράγραφο ακριβώς για αυτό το θέμα. That'll be it. That'll be it for this. Αυτά είναι. Τελειώσαμε αυτό το σημείο της ημέρας της διάταξης. Οπότε μπορούμε να πάμε παρακάτω στο θέμα που αφορά την Ευρωπαϊκή Φυλακή και Ακτοφυλακή. Ευχαριστώ για όσου ήρθαν, χωρί να είναι τακτικά μέλη και ήρθαν για να συμμετάσχουν στη συζήτηση του προηγουμένου θέματο και τώρα φεύγουν. Αλλά παρακαλώ προσέξτε γιατί πάμε στο επόμενο θέμα, συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή. Από ό,τι μου λένε όμως, η εισηγήτρια, κυρία Μετσόλα, ε, οφείλει να είναι εδώ σε ένα λεπτό. So if I, uh, may require your patience, let's wait an additional minute. Να επιδείξετε υπομονή να περιμένουμε αυτό το λεπτάκι. Ούτως ώστε να έρθει η κυρία Μετσόλα και να αρχίσουμε. Είναι η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 Ευχαριστώ για την υπομονή σας, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα που έχει έρθει η συγγήτρια, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι την περσμένη εβδομάδα είχαμε τον εκτελεστικό διευθυντή την Frontex που μας ε, ενημέρωσε για τις δραστηριότητε της υπηρεσίας και συζητήσαμε τα της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Frontex. Σήμερα θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεσης για συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή. Κύριε Μετζόλα, η συνάδελφος είναι η συγγήτρια και της δίνω τον λόγο. Πέντε λεπτά. Και μετά θα συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δουλέψαμε εντατικά τις τελευταίες εβδομάδες για να συντάξουμε αυτή την έκθεση και καταλήξαμε στις προτάσεις μας για το ποιος είναι ο πιο ρεαλιστικός και αποτελεσματικός τρόπος ε, που πρέπει να προχωρήσει η υπηρεσία. Να μην ε, δούμε μία-μία τις τροπολογίες. Απλώ ε, απλώς περιμένω να ακούσω την αρχική εντύπωση των συναδέλφων μου και βασική αλλαγή της Επιτροπής είναι η, ο πυρήνας της δραστηριότητας της ε, υπηρεσίας. Όλοι ξέρουν ποια είναι τα δυνατά σημεία στην υπηρεσία αυτή και το τι πρέπει να γίνει για να μπορεί να αναπτυχθεί όπως πρέπει αυτή η υπηρεσία στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρχει πάντως ε, ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, έχουν προκύψει πάρα πολλά ερωτηματικά και στα μέσα ενημέρωσης και στα άλλα θεσμικά όργανα. Οπότε για αυτό και εγώ θα πρέπει να υπάρχει μια τέταρτη κατηγορία προσωπικού. Να υπάρχει ε, αυτό το προσωπικό των τριών χιλιάδων που να χρησιμοποιούνται σαν ταχεία δύναμη αντίδραση όταν υπάρχει κάτι το έκτακτο το κατεπήγον. Να δούμε πώς θα πλαισιώσουμε τις κατηγορίες 1 έως 3 να έχουμε 30% να μην υπάρχει το, το, το κατόφλι αλλά να έχουμε 5 έως 20.000 ε, άνω και κάτω όρια για το προσωπικό και όλα αυτά να ισχύσουν πέντε χρόνια μετά τη θέση ισχύ του κανονισμού. Και βέβαια αυτά σας τα λέω αφού πήρα τη γνώμη κάποιων που ασχολούνται στην πράξη με το θέμα. Γιατί στις επιστροφές θα πρέπει αυτές οι, αυτοί οι επαναπατρισμοί να γίνονται με κάθε εγγύηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να έχουμε κάποιες ρήτρες διασφάλισης που να δεσμεύουν την υπηρεσία σε σχέση με μετακινήσεις από τρίτη σε τρίτη χώρα. Και κάθε διαπραγμάτευση θα πρέπει να γίνεται επί τη βάση κάποιας προηγουμένης αξιολόγησης και κοινοποίηση στο Κοινοβούλιο σχετικά. Πέραν αυτής της αξιολόγησης να έχουμε συγκεκριμένη αξιολόγηση το τι γίνεται με την τρίτη χώρα και τις, τους επαναπατρισμούς ε, και επίσης για ε, μετακινήσεις από τρίτη χώρα σε άλλη τρίτη χώρα. Οπότε θα πρέπει η πανέβαση να γίνεται ε, σε χώρες και περιοχές ε, που θεωρούνται από τον ΟΗΕ ασφαλής. Θα πρέπει να δούμε με τους κοιοδησηγητές πως ε, όλα αυτά θα συμβάλλουν στην πράξη σε εύρυθμη λειτουργία. Βασικά σε όσα μου είπαν οι συνάδελφοι και ήθελα να θωρακίσω τον μηχανισμό καταγγελιών και τον υπάλληλο που ασχολείται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, εγώ σε επαφή με πολλούς εμπλεκομένους και ανέδειξα τα προβλήματα που επιτόπου διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν στα σύνορα, τα εξωτερικά και το πρόβλημα είναι η έλλειψη σε ανθρώπινους πόρους και χρηματικούς πόρους. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη ε, αυτόν τον πυρήνα της υπηρεσίας να κρυθεί. Ακριβώς τι θα έχει το προσωπικό της υπηρεσίας για το θα πρέπει να φέρουν όπλα όταν γίνεται κάποια επιχείρηση και ως εκτελεστική αρμοδιότητα να δούμε το τι θα γίνει με τις θεωρήσεις. Αυτό θα πρέπει να γίνεται μόνο από εθνικούς υπαλλήλου, γιατί εδώ θα πρέπει να κατησχίσει η επικουρικότητα. Τώρα για άλλες ε, τροποποίησεις που προτείνω είναι η εκπαίδευση και θέλω να υπάρχει ένας μηχανισμός ε, ελέγχου ποιότητας και εξωτερικός έλεγχος επίσης για όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης. Θα πρέπει να δούμε ανατομέα πώς θα γίνει η διαχείριση των συνόρων και οπότε η, αυτά τα οριζόντια συστατικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη να αναβαθμιστεί ρόλο του Κοινοβουλίου για κάθε θέμα του κανονισμού. Επέλεξα το να συνεχιστεί αυτό που συμφωνήθηκε μεταξύ των συνομοθετών δύο χρόνια πριν. Δεν λέω εδώ πέρα τίποτα το, τόσο καινούριο. Οι ανάγκε ανάγκες τώρα στα κρατημέλη που έχουν κάποια διάρκεια και σε τροπολογίες λέω ότι θα πρέπει οι υπηρεσίες που φροντίζουν για αυτά τα πυρητσακά καθήκοντα να υπάρχουν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου κάνουμε επιστροφές, επαναπατρισμούς και βέβαια και προκειμένου να υπάρχει λογοδοσία και κοινοβουλευτικός έλεγχος. Βλέπετε ότι το θέμα έχει μεγάλη εμβέλεια. Περιμένω πώς και πώς να ακούσω συναδέλφους, αλλά και τους κοιόδης εισηγητές για το πώς βλέπουν τις προτάσεις μου. Και όλα αυτά εν ώψη του χρονοδιαγράμματος για τις τροπολογίες. Και θέλω τελικά να καταλήξουμε σε μια συνετική λύση που να συμφωνούν όσο γίνονται περισσότερε πολιτικές ομάδες. Σας ευχαριστούμε κυρία Μετσόλα. Αυτή είναι η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης. Ήρθε η ώρα των σκιωδών εισηγητών. Ο κύριος Σίντερ είναι ο πρώτος σκιώδης εισηγητής που θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα θυμάστε ότι το 2016 οι συνομοθέτες κατάφεραν να υιοθετήσουν ε, γρήγορα τον κανονισμό για το Frontex με θέση ισχύ αργότερα στο ίδιο έτος. Και μάλιστα ο εφαρμοστικό κανονισμό μετέτρεψε το Frontex σε ένα πλήρη οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διευρυμένη εντολή. Δύο χρόνια αργότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταθέτει μια άλλη πρόταση για την ενίσχυση, περαιτέρω ενίσχυση της εντολής του Frontex. Ευχαριστώ την κυρία Μετσόλα για το πολύ αξιόλογο έργο της, γιατί το σχέδιο έκθεσης ε, τηρεί πιστά το πνεύμα της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, γι' αυτό θα το εξετάσω πολύ προσεκτικά. Η έκθεση όμως περιλαμβάνει κάποια στοιχεία που επίσης με βρίσκουν σύμφωνο, όπως ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η επικέντρωση στην ε, επιμόρφωση και κατάρτιση και φυσικά συμφωνώ και με την ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά το μόνιμο σώμα του Frontex, πολύ ρεαλιστική έκθεση, αξιοποιώντας ε, ήδη το προσωπικό των 1500 ε, μελών της ομάδας ταχείας αντίδρασης. Και σίγουρα σημαντικό θέμα είναι η συμμετοχή του Frontex σε επιστροφές από και προς τρίτες χώρες. Δεν είμαι πεπισμένος για την ε, ανάγκη ε, θέσπιση τέτοιων διατάξεων ούτε το 2016 ούτε και τώρα. Κατά τη γνώμη μου αυτό περισσότερο έχει σχέση με τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι με τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων η εκχώρηση εκτελεστικών εξουσιών στα μέλη του Μονίμου Σώματος για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων ε, του Frontex είναι κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί με μεγαλύτερη προσοχή. Τα μέλη θα ακολουθούν τι εντολέ των ενδιαφερομένων κρατών μέλων. Αυτό όμω σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη θα είναι υπεύθυνα για τι δράσει του οργανισμού αυτού. Κατά τη γνώμη μου, η ενίσχυση της εντολής του οργανισμού θα πρέπει να συνοδευτεί με ενίσχυση της λογοδοσίας και της ευθύνης του οργανισμού. Χρειάζεται υποπτία ε, σε όλες τις δραστηριότητες ε, του Frontex, ιδιαίτερα στις επιστροφές, αλλά και στο διορισμό του εκτελεστικού διευθυντή και των, των αναπληρωτών εκτελεστικών διευθυντών. Τέλος, ε, η ομάδα μου είναι έτοιμη για στενή και επικοδομητική συνεργασία με την κυρία Μετσόλα γιατί θεωρούμε ότι η έκθεσή τη είναι πολύ σημαντική και ω εκ τούτου οι σοσιαλιστέ και οι δημοκράτε θα είναι όσο πιο επικοδομητικοί γίνονται στην ε, διαδικασία των συζητήσεων με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ κύριε Νίδερ Μίλλερ. Εκ μέρου ε, των συντηρητικών μεταρρυθμιστών ο κύριο Βίστικεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κατάλαβα ότι εννοούσατε εμένα. Κανένα πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Εισηγήτρια, σας ευχαριστούμε για το σχέδιο του εγγράφου εργασία σας για να έχουμε μια βάση για τις διαπραγματεύσεις μας. Γενικώ είμαι υπέρ ε, του, του νέου οργανισμού συνοριακής και εκτοφυλακής ε, για να ελέγχουμε την κίνηση εξωτερικά μας σύνορα που σημαίνει ε, ότι ο έλεγχος των εξωτερικών σύνορων είναι κοινή συλλογική ευθύνη όλων των κρατών μελών και θα πρέπει να ε, ληφθεί όντω υπόψη. Η κρίση έχει εκθέσει κατάφορα τις περίτρανα μάλλον τις αδυναμίες και τα κενά που υπάρχουν στους ε, τρέχοντες μηχανισμούς. Και για να ξεπεράσουμε αυτά τα κενά και τις αδυναμίες, πιστεύω ότι ο οργανισμός ε, συνοριοφυλακής και εκτοφυλακής θα διδραματίσει και ρόλο. Είμαι υπέρ αύξηση του προσωπικού και του εξοπλισμού, είμαι υπέρ της ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων, για την επιστροφή των των που έχουν απορριφθεί αιτήσει τους στις χώρες και μεγαλύτερη συνεργασία και η συμπερίληψη του Eurosur ε, στη λειτουργία του οργανισμού. Δεν βλέπω ότι έχει λόγο να προσθέσουμε νέε αρμοδιότητες ή να μεταφερθούν αρμοδιότητες ε, για τις πολιτικές ε, που καθοδηγούν τον οργανισμό. Και σίγουρα ε, δεν θα πρέπει να γίνει μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Συμβούλιο στην Επιτροπή, ιδιαίτερα σε έκτακτες περιστάσεις. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, κρατούν αυτές τις ευθύνες και να αναλάβουν ε, τις ευθύνες των δράσεών τους. Βέβαια, αναφέρθηκαν κάποιες επιφυλάξεις για την ανάπτυξη του οργανισμού σε τρίτες χώρες, την αύξηση του προσωπικού και την ενίσχυση τη της εντολής της ό,τι αφορά τις επιστροφές. Αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες κάποιου συναδέλφου για τα θέματα αυτά και προσβλέπω σε περαιτέρω επικοδομητική συνεργασία με την εισηγήτρια. Σας ευχαριστώ που μου δώσετε το λόγο. Μάλιστα, εκ μέρου των φιλελευθέρων, ο κύριος Ντεπχέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αντικαθιστώ τη συνάδελφο Ναταλή Γκρισπέκ, που ζητά συγγνώμη για την απουσία της. Επιτρέψτε μου λοιπόν να διαβάσω τις προτάσεις της κυρίας Γκρισπέκ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τη ρησηγήτρια Ρομπέρτα Μοτσόλα, που πραγματικά ε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα επιτέλεσε πραγματικά ένα πολύ αξιόλογο και άρτιο έργο. Η κυρία Μετσόλα ε, κατέδειξε πολύ σημαντικά θέματα σε ό,τι αφορά το μόνιμο προσωπικό, τις εκτελεστικές ε, εξουσίες, αλλά και τα μισθολογικά ζητήματα του νέου οργανισμού. Ε, μάλιστα ενισχύονται κάποιες διατάξεις που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα, το σεβασμό τους και προτίζει την σύσταση μιας μονάδας ε, εποπτείας. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση της κυρίας Μετσόλα. Επίσης είμαι υπέρ της ενίσχυσης και της εξασφάλισης της ανεξαρτησίας του υπαλλήλου του αρμόδιου για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει οι αρμόδιοι υπάλληλοι να έχουν όλες τους πόρους, τα εφόδια και το χρόνο για να διεκπαιρεώσουν σωστά το έργο τους. Κατά τη γνώμη μου, η στόχη είναι η εξή. Ό,τι αφορά το μόνιμο προσωπικό, διαρωτώ με αν είναι εφικτή η παρούσα πρόταση που ζητάει ένα μόνιμο σώμα 10.000 υπαλλήλων μέχρι το 2020. Θα είναι πολύ δύσκολο να στελεχωθεί ένα τέτοιο σώμα. Θέλουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα στις προθεσμίες. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την κατάρτιση, την επιμόρφωση, η κυρία Μετζόλα ενίσχυσε τις διατάξεις για τα θέματα κατάρτισης. Η κυρία Γκρισμπέκ όμως θα ήθελε ο ίδιος ο οργανισμός ε, να εκπαιδεύει τους συνοριοφύλακες και τους ε, ακτοφύλακες ε, του σώματος. Αν θέλουμε πραγματικά μια πραγματική παιδεία εντός του οργανισμού, μια κουλτούρα του οργανισμού, θα πρέπει ο οργανισμός να εκπαιδεύει και να καταρτίζει τις ομάδες του. Επίσης θα πρέπει να διευκρινιστεί το κείμενο της πρώτης κανονισμού, αλλά είναι πολύ περίπλοκο το σχετικό, ε, το σχετικό τμήμα. Για παράδειγμα, εκτελεστικές εξουσίες ή πρόσβαση στα δεδομένα τι δικαιούνται ή τι δεν δικαιούνται να κάνουν οι υπάλληλοι του Frontex, του νέου οργανισμού. Θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Είναι πολύ συγκεχημένα τα πράγματα αυτά. Επίσης κάτι που είναι πολύ συζητήσιμο και θα συζητηθεί όντω, δυνατότητα πραγματοποίηση επιστροφών από μία τρίτη χώρα σε άλλη, από τον ίδιο τον οργανισμό. Αυτό το ζήτημα και εμένα με προβληματίζει όπως και πολλούς συναδέλφους. Τέλος, κάποια άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα ακούσαμε κάποια πολύ σημαντικά σχόλια στην Επιτροπή Λύπε, από τον Διευθυντή του Οργανισμού, τον Φαμπρίς Ζέρι. Η διαχείριση των συνόρων, είπε, δεν σημαίνει διαχείριση μόνο των μεταναστευτικών ροών, αλλά και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι μαζί πώς θα δώσουμε έμφαση σε αυτά τα στοιχεία. Αυτές είναι σε γενικές γραμμές οι θέσεις των φιλελευθέρων εκ μέρους της τη ηγετρίας, η οποία θα καταθέσει εμπρόθεσμα και τροπολογίες. Ευχαριστώ και πάλι την κυρία Ρομπέρτα Μετσόλα, την εισηγήτρια, που επαναλαμβάνω επιτελεί ένα πολύ αξιόλογο έργο και την ευχαριστώ γιατί αφογκράστηκε ιδιαίτερο στις θέσεις των συναδέλφων. Αυτέ είναι οι απόψει τη κέντρου ηγετρία των φιλελευθέρων, κυρία κυρίας Γκρισμπέκ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντεπρέ. Η κυρία Γκόμε. Ε, θέλετε να πάρετε το λόγο να κάνετε σχόλια. Then... Ζητώ συγγνώμη. Να ακούσουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν επισημαίνει πάρει το λόγο. Πρώτος δώσουμε το λόγο και πάλι στην εισηγήτρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ και καλησπέρα σα. Δεν έχω πολλά να προσθέσω στην παρούσα φάση. Διαβάσαμε με προσοχή και ενδιαφέρον την έκθεση. Χαιρόμαστε που καταρτίστηκε τόσο γρήγορα. Είναι πολύ υψηλής ποιότητος. Στην παρούσα φάση, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να σχολιάσει τις προτινόμενες ε, τροπολογίες σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο. Ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας. Μάλιστα. Θέλετε να πάρετε το λόγο για να κλείσετε τη συζήτηση, κυρία Μέτσολα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και θα μιλήσω στην δική μου γλώσσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους ε, που πήραν το λόγο ήταν πολύ θετική και χαίρομαι γι' αυτό. Να απαντήσω σε κάποια από τα ζητήματα τα οποία θίξαν οι συνάδελφοι σε ό,τι αφορά ε, τις εκτελεστικές αρμοδιότητες. Προσπαθώ λοιπόν να δω τις ε, περιορισμούς που υπάρχουν προκειμένου να διευκρινιστεί ότι το κράτος μέλος υποδοχής είναι αυτό που θα χορηγήσει τις εκτελεστικές αρμοδιότητες και θα πρέπει να δράσει. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των 10.000 μέχρι το 2020, αναγνωρίζω το χρονικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ήταν πολύ φιλόδοξο. Και μετά από συνομιλίες με διάφορους κυβερνητικούς εκπροσώπους, καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει να παραταθεί αυτό το χρονικό όριο. Σε ό,τι αφορά τώρα την Ακαδημία Εκπαίδευση, από αυτά που είπε η συνάδελφο η κυρία Γκρίσπεκ, καταλαβαίνω τη θέση τη. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι θα πιστεύει ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η νοοτροπία στον Frontex, ότι όλοι θα πρέπει να έχουν την ίδια εκπαίδευση, όλοι που απασχολούνται στο Frontex. Υπάρχουν επίσης κάποιες δυσκολίες, ε, γιατί ενδεχομένως να ανεβάσει το κόστος εκπαίδευσης αυτό. σε ό,τι αφορά και την προσέλκυση εκπαιδευτών, οι οποίοι προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Αλλά θα δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την κατάσταση αυτή σε ό,τι αφορά το κείμενο για το οργανωμένο έγκλημα. Πιστεύουμε ότι ενδεχομένως να ενισχύσουμε τις δομές αυτές και περισσότερο από ό,τι αναφέρω. Επίσης, Ε, εισηγάγαμε αυτούς τους πέντε περιορισμούς ε, και ενδεχομένως αυτό να μας οδηγήσει σε, μια, ένα κατάλογο χωρών. Συναντηθήκαμε με τον κύριο Λετζέρη, ο οποίος και μας είπε ότι θα ήθελε να υπάρχει δυνατότητα επιστροφής, αιτήματος για επιστροφή επικόντρα της χώρας ε, με ασφαλείς όρους. Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι η κατάσταση αυτή ενδεχομένως να παρουσιαστεί και σε γειτονικέ χώρες. Όταν θα φτάσουμε στο σημείο που θα κατατεθούν τροπολογίες, θα δω πώς θα μπορούσα να καταθέσω και μια συμβαστική πρόταση. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μέτσολα. Κανείς άλλος στο θέμα αυτό? Να περάσουμε στο τελευταίο πακέτο, της θεωρήσης. Εγώ είμαι ο εισηγητής, αν μου επιτρέψετε. Οπότε τώρα θα έχω το διπλό ρόλο του Πρόεδρου και του εισηγητή και θα κάνω την παρουσίαση του θέματος. Πρώτα-πρώτα αυτά είναι το σημείο παριθμών 8 που αφορά την ε, συζήτηση των τροπολογιών για τον ενωσιακό κώδικα κώδικα ο οποίο προβλέπει κάποιε προποθέσει, κάποιε διαδικασίε για την έκδοση θεωρήσεων διαβατηρίων για σύντομη διαμονή και ε, διάβαση από τα, ε, από τα αεροδρόμια. Είναι πρόκειται 284 τροπολογίε. και επιτρέψτε μου να σα ε, πω τα τη έκθεσή μου όσον αφορά τι τροπολογίε και στη συνέχεια να συνδυάσουν το θέμα αυτό με το 9 και εκεί είμαι εισηγητή και αφορά τις θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους. Να δούμε τώρα τις τροπολογίες όσον αφορά αυτόν τον κώδικα ε, θεωρήσεων. Όπως σας προανέφερα, ε, έχουν υποβληθεί αρκετές ε, τροπολογίες για την έκθεση. 174 της ΓΚΟΕ. Ε, περίπου 30 της ΓΚΟΕ, των Πρασίνων, 14 από το ΕΡΑΚ και μερικές από τη δική μου πολιτική ομάδα και έχουμε και 20 από το ENF. Καμία από το ECR, άρα το ECR είναι ικανοποιημένο από την πρόταση της Επιτροπής. Οι περισσότερες αυτές τις τροπολογίες προέρχονται από το Elk και την ALDE. Είναι τεχνικές και αφορά ε, τεχνικά χαρακτηριστικά, λειτουργία αυτού του κώδικα. Η Πράσινη και η ΓΟΕ ε, υπέβαλαν πιο γενικόλογες τροπολογίες πολιτικού χαρακτήρα. Ορισμένε από αυτέ έχουν και τεχνικό χαρακτήρα, αλλά πολλέ θέλουν να ενισχύσουν την ανθρωπιστική διάσταση του κώδικα θεωρήσεων. Σκληρά δουλέψαμε με τους σκιώδεις εισηγητές για να καταλήξουμε σε συμβαστικέ τροπολογίες και προσπαθήσαμε να δουλέψουμε ταχύως γιατί θέλουμε στις 3 Δεκεμβρίου στην Λίμπε να γίνει η ψηφοφορία αυτό χρειάζεται εάν θελήσουμε να έχουμε έγκριση του έκθεση πριν το τέλος της ε, θητείας που πλησιάζει, δεν έχουμε και τόσο χρόνο να μας απομένει. Επίσης, περί τον Φεβρουάριο έχουμε άλλα θέματα που αφορούν αυτή την τελική ευθεία αυτής της θητείας. Να κάνουμε επομένως ό,τι μπορούμε για την υπόθεση αυτή. Παρακαλώ βοηθήστε με να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Βέβαια δεν μπορούσαμε να φτιάξουμε συμβαστικές για όλες τις τροπολογίες γιατί πολλές φορές υπήρχαν τόσες ε, αντιφάσεις, τόσες αντιθέσεις που δεν άφηναν περιθώριο για συμβασμό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα γίνουν χωριστά οι ψηφοφορίες για τις εν λόγω τροπολογίες. Και τώρα, για να πούμε για ε, τις βασικές τροπολογίες ανά θεματική ομάδα. Πρώτα πρώτα αυτές που αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την έκδοση θεώρησης. Ιδίω όσον αφορά αθλητισμό και πολιτιστικά. Ε, Γκουε και ΕΛΚ και νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση υπέρ αυτών των τροπολογιών. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ένα μια άλλη ενότητα όσον αφορά ιατρικό ταξίδι. Η διευκόλυνση είναι λογική, λένε οι περισσότερες πολιτικές ομάδες. Τρίτη κατηγορία προτάσεων και τροπολογιών όσον αφορά ε, το κόστος της ε, θεώρησης. Και εδώ έχουμε τροπολογίες προς πάσα κατεύθυνση. Κάποιοι θα θέλανε να είναι το σχετικό τέλος τα σχετικά έξοδα λιγότερα. Άλλοι θέλουν να ανέβει η σχετική τιμή. Άλλοι θέλουν να συνδεθούν ε, τα έξοδα με την οργάνωση της κοινότητα, με την οικογένεια, με την ηλικία του ετούντος εμείς. Δουλεύουμε σκληρά να βρούμε μια συμβαστική για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις διαστάσεις για τα έξοδα. Και υπάρχουν κάποιες θετικές προτάσεις από τον κύριο Ντεπρέ θα τα λάβουμε υπόψη για να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Και όπως είπαμε πριν, στην πρώτη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών, προσπαθούμε να δούμε τα τεχνικά σημεία και με... η τροπολογία 21 θέλω να καταλήξω σε συμβιβασμό όσον αφορά τα έξοδα ε, των θεωρήσεων. Τώρα είδα και τις δικές σας ε, τροπολογίες και έχω την τροπολογία 23 και την 163 του κυρίου Ντεπρέ. Αυτές οι τροπολογίες είναι συμβατές και αυτές θα πρέπει να είναι ε, η βάση μιας συμβαστικής τροπολογίας για το άρθρο 17, παραγραφός 4, αυτού είδους το τέλος, το, το service fee, το τέλος εξυπηρέτηση, θα πρέπει να καλύπτει τα πάντα. Ο, ο κάθε κόστος που έχει σχέση με την αίτηση για απόκτηση θεώρησης. Θα πρέπει ο κόσμος τον προτέρων να ξέρει πώς θα του κοστίσει η θεώρηση πριν υποβάλει την αίτηση. Και εδώ υπάρχουν διάφορα στοιχεία για συμβαστικό και καλύπτουμε την τροπολογία του κυρίου Ντεπρέ που είπαμε ότι θα είναι βάση συμβασμού με όλους τους σκιώδες. Τώρα, ε, πέμπτο σημαντικός κύκλος είναι για την έκδοση ομοιόμορφης θεώρησης άρθρο 24. Εδώ είναι αυτό το ε, σύστημα ε, Accepting the Commission proposal for accessing the first visa. Δηλαδή, για ένα κύμα από θεωρήσεις. Δηλαδή, να δίνεται η πρώτη και μετά να διευκολύνεται η χορήγηση των υπολείπων. 194 πρώτη κύριο Δεπρέ και την 193. Ε, οι υπόλοιπες τροπολογίες για αυτό το άρθρο παρακαλώ στηρίξτε την τροπολογία με αριθμό 32. Δύσκολο να βρούμε τροπολογία, έχουμε και άλλες. Ιδάλλως θα πρέπει να γίνει πάλι στην ψηφορία. Έκτο η θεματική ενότητα αφορά τους κινδύνους προς ασφάλειας και μετανάστευσης. Προσωπικά και πολύ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να πάμε προς τα εκεί, γιατί υπάρχουν πολλές διασφαλίσεις. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει γνωστή ψηφορία όσον αφορά αυτά τα σημεία δεν συμφωνείτε με τη δική μου πρόταση, δηλαδή ότι θα πρέπει ε, αυτή η διάταξη να διαγραφεί για αυτούς τους κινδύνους. Θεωρώ ότι αυτό το βρίσκει σύμφωνη την κυρία Βερζιάτ και την κυρία Βαλέρο. Επίσης το άρθρο 25, τη σχέση με την επανεισδοχή. Για πολλές πολιτικές ομάδες Εδώ θα πρέπει να διευκολύνεται η συνεργασία με τις τρίτες χώρες για την επανεισδοχή. Ξέρετε ότι αυτή η λογική με βρίσκει πολύ αντίθετο. Άρα δεν θέλω να καλύψουμε τέτοια προσέγγιση της ε, Επιτροπής. Όμως σε πολλές συναντήσεις που ήδη κάναμε για το θέμα και εν ώψη ε, των ε, διαφορετικών τροπολογιών μέχρι τώρα θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια διασύνδεση των θεμάτων, να βρούμε δηλαδή συμβαστική τροπολογία και έτσι να βρούμε την ισορροπία. Στο μέτρο του δυνατού. Ε, και εδώ έχουμε πρόταση του κυρίου Ντεπρέ, να υιοθετηθεί ένα σύστημα που να προβλέπει κάποιο είδους κίνητρα, θετικά κίνητρα, για τις χώρες που θέλουν, για την ε, επανεισδοχή να συνεργαστούν. Όχι μόνο για τις αρνητικές συνέπειες, αλλά να υπάρξει ισορροπία μεταξύ αυτών των θετικών κινήτρων και της διασύνδεσης με την υπόθεση της επανεισδοχής. Αυτό είναι βάση για συμβαστική τροπολογία, για συμβασμό. Τέλος, για την ανθρωπιστική διάσταση των θεωρήσεων. Ξέρετε ότι για μένα είναι σημαντικό το ότι παρετήθηκα από τον έχουμε στον κώδικα των θεωρήσεων τέτοιο θέμα, τέτοια αμνία. Όλα αυτά λόγω τη αντίθεση θέση του Συμβουλίου η Επιτροπή και κάποιες πολιτικές ομάδες εδώ επίσης ήταν αντίθετοι και τελικά είπαμε ότι μόνη διέξοδο είναι να προωθηθεί αυτή η πρόταση με την έκθεσή μας ιδέες πρωτοβουλίες για τις ανθρωπιστικές βίζες. Οπότε θα σας τα πω. Στα πλαίσια εκείνης έκθεσης μετά από την τωρινή συζήτηση για τον κώδικα θεωρήσεων. Είπαμε, θα κινηθεί παράλληλα η εκθεσία της πρωτοβουλίας για τις ε, ανθρωπιστικές θεωρήσεις, παράλληλα με αυτήν την έκθεση. Ελπίζω ότι στις 3 θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας, κατόπιν θα εγκρίνει η Ολομέλεια το θέμα. Οπότε και θα έχουμε χρόνο να ολοκληρώσουμε κατά αυτή την ε, χρονιά. Πριν τις χρονιάτικες διακοπές. Ε, και εννοείται οπωσδήποτε πριν το τέλος της θητείας. Αυτό θα ήταν το ιδιώδες. Ανέκαθεν θεώρησα ότι η πολιτική των θεωρήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναδείξει το πόσο είμαστε δεσμευμένοι ε, όσον αφορά τι, τι δράση θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω, τι εικόνα. Και γι' αυτό και πρότεινα κάποιες τροπολογίες για να ενισχύσω αυτή την πλευρά του θέματος και οι κυρίες Βαλέρο και Βερζιάτ έκαναν το ίδιο και νομίζω ότι κάποια από όσα πρότειναν μπορούμε να τα καλύψουμε στο κείμενο. Εάν δεν μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβασμό, αυτές οι τροπολογίες θα ψηφιστούν χωριστά και εκείνες. Πάντως ελπίζω ότι η πλειοψηφία εξημών καταλαβαίνει ότι θα πρέπει αυτή η ανθρωπιστική διάσταση να παραμείνει και να εγκρίνουν την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. για την ανθρωπιστική θεώρηση που θα συζητήσουμε μετά. Τώρα να ακούσουμε τη γνώμη των ε, σχεδόν συγκεκριτών. Κύριε Μπέικερ, εσείς πρώτος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και νομίζω ότι είναι πολύ σκόπιμο να προσπαθήσουμε το θέμα αυτό του κώδικα θεωρήσεων να το ολοκληρώσουμε πριν από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, πριν από την αλλαγή του έτους. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις προσπάθειες που κατέβαλε και τους σκιώδες εισηγητές που προσπάθησαν να διαμορφώσουν συμβιβαστικές προτάσεις. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στο εξή ε, σημείο η συνεργασία με τα τρίτα κράτη, με θέλουμε να είναι βέλτιστη. Γιατί εδώ μιλάμε για επιχειρηματίες, για αθλητές, για καλλιτέχνες και τουρίστες. Θέλουμε λοιπόν να καταστεί πιο εύκολο για αυτούς να ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Και άρα θέλουμε κάποια απλοποίηση σε ό,τι αφορά την έκδοση θεωρήσεων. Πέραν τούτου, θα πρέπει να δημιουργηθούν μοχλοί σε ό,τι αφορά τις θεωρήσεις που θα υποστηρίξουν τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά τις ε, επιστροφές και εξ ονόματος της πολιτικής μας ομάδας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αυτή η πολιτική θεωρήσεων που έχει ως βάση την επανειστοχή είναι πολύ σημαντική για μας. Θέλουμε να υπάρχει επικοδομητική σχέση με τα, κράτη, με τα άλλα κράτη. Θα πρέπει να είναι εύκολο λοιπόν να αποκτήσουν θεωρήσεις ε, οι υπήκοοι των χώρων αυτών, εφόσον τα πράγματα λειτουργούν σωστά. Εάν δεν λειτουργούν σωστά, θα πρέπει να υπάρξουν συνέπειες. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Βλέπουμε λοιπόν στην έκθεση στοιχεία τα οποία δεν μπορούμε να τα υποστηρίξουμε ολοκληρωτικά στην παρούσα φάση σε ό,τι αφορά για παράδειγμα η διευκρινήση του πώς θα μπορούσαν να αποκτήσουν οι αθλητές πρόσβαση σε τέτοιες θεωρήσεις και κυρίως ε, θεωρούμε ότι δεν είναι, παραδεκτή, δεν είναι αποδεκτή η ρήτρα για την επανένωση οικογενειών. Σε ό,τι αφορά επίσης ε, τους ασθενείς, εδώ θα μπορούσαμε να δεχτούμε κάποια μέση λύση και να κατατεθούν αμ, τροπολογίες. Σε ό,τι αφορά το τέλος έκδοσης ε, της θεώρησης, θεωρούμε ότι θα πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον ε, ο συντελεστής του πληθωρισμού. Αυτό δεν γίνεται στην παρούσα φάση. Δεν καλύπτονται λοιπόν τα έξοδα στην παρούσα φάση με τα προτινόμενα τέλη. και είναι ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο πολύ καλή η τιμή έκδοσης των θεωρήσεων. Όποιος δεν μπορεί να πληρώσει μία θεώρηση στα πλαίσια του χώρου Σέγγεν, δεν θα μπορέσει έτσι κι αλλιώς να κάνει σπουδαία πράγματα στην Ευρώπη, γιατί τα έξοδα διαβίωσης στην Ευρώπη είναι πολύ πιο υψηλά από την έκδοση της ε, θεώρησης. Σε ό,τι αφορά τη διευκρίνηση για τα μέλη ΜΚΟ κατά των 30 ετών, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό που προτείνεται. Γιατί στην τελική ανάλυση πιστεύουμε ότι αν ισχύει κάτι τέτοιο, όλοι οι υπήκοοι των χωρών θα ήταν μέλη κάποια ΜΚΟ. Αυτό δεν έχει νόημα. Η διαγραφή τώρα του τμήματος για τη μετανάστευση, αν μπλοκ στην έκθεση, είναι κάτι που δεν το αποδεχόμαστε. Και γι' αυτό ε, ο εισηγητής νομίζω ότι θα έπρεπε να προτείνει μια ονομαστική ψηφοφορία για τα θέματα αυτά γιατί θα πρέπει να ξέρουμε ποιος ε, λέει λατή αυτά τα δύο σημαντικά ζητήματα για τους πολίτες. Και επίσης πιστεύουμε ότι τίθεται θέμα κινδύνου ή ασφάλεια. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε διάφορα σημεία σε ό,τι αφορά την ασφάλεια. Αλλά θέλουμε να είναι σαφώς διατυπωμένες οι συμβαστικές προτάσεις. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Και αν ε, υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις, θα συμφωνήσει και το ΕΛΚ και θα υπερψηφίσει την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. ευχαριστούμε κύριε Μπέκερ. Κυρία Στίβενς τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και συνάδελφοι. Θα ήθελα, όπως και προηγουμένως ε, ομιλητής, να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τις κοιότητες εισηγητές για την συνεργασία τους σε ένα τέτοιο σημαντικό θέμα. Σημειώσουμε κάποια σημαντική πρόοδο, διαπιστώνω, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε να προωθήσουμε τον τουρισμό μας, να μπορούμε να πείσουμε τον κόσμο να επισκέφτεται την Ευρώπη. Και χρειαζόμαστε λοιπόν ε, σαφείς ε, κανόνες και ομοιογενείς ε, κανόνες για τις θεωρήσεις και για τους επιχειρηματίες, τους μουσικούς, καλλιτέχνες, performers, όλα αυτά λοιπόν συμπεριλαμβάνονται. Όπως ανέφερε και η πολιτική ομάδα του ΕΛΚ και εμείς έχουμε από την πολιτική μας ομάδα προτάσεις σε ό,τι αφορά το κείμενο του εισηγητή. Συνολικά θέλουμε να παραμείνουμε αρκετά κοντά στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορούμε να υποστηρίξουμε κάποιες ε, τροπολογίες, κάποιες άλλες δεν θα μπορέσουμε να τις υποστηρίξουμε σε ό,τι αφορά για παράδειγμα τους αθλητές ε, και καλλιτέχνες ε τραγουδιστές και ούτω καθεξής. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουν τους ίδιους όρους ό,τι αφορά την έκδοση θεώρησης όπως όλοι οι υπόλοιποι. Είναι σημαντικό αυτό. Σε ό,τι αφορά τις ιατρικές ασφάλειες για ταξίδι, δεν είμαστε υπέρ της διαγραφής αυτών. Όταν ένα άτομο είναι ασθενής, ε, αυτό συνεπάγεται συγκεκριμένο κόστος. Δεν μπορούμε λοιπόν να αφήσουμε τον ασθενή να επομιστεί όλο αυτό το κόστος. Θα πρέπει να έχει δυνατότητα να ασφαλίζεται σε περίπτωση ασθένειας. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται η θεώρηση για τους ασθενείς. Σε ό,τι αφορά το κόστος, το τέλος για την έκδοση των θεωρήσεων, υποστηρίζουμε την προτινόμενη τιμή για το τέλος αυτός, γιατί θεωρούμε ότι αυτό καλύπτει λίγο πολύ όλα τα έξοδα που συνδέονται με την έκδοση της θεώρησης και παραμένουμε φυσικά ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να εξεταστούν κάποιες ε, εκπτώσεις ε, για κάποιες ομάδες ε, του πληθυσμού, για παράδειγμα για τους ανήλικους. Εξωτερική ανάθεση τώρα. Πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να φορτωθούμε το κόστος της εξωτερικής ανάθεσης. Όσοι θέλουν να το αναλάβουν θα πρέπει να αναλάβουν και το κόστος. Σε ό,τι αφορά τις ε, διατάξεις ε, για τις θεωρήσεις ε, και τις επιστροφές. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντική αυτή η σύνδεση. Είναι σημαντικός αυτός ο σύνδεσμος. Αν μια χώρα θέλει να έχει πρόσβαση σε τέτοια διευκόλυνση για θεωρήσεις, θα πρέπει να συνεργάζεται για πιο πολλές επιστροφές. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα δύο να είναι αλληλοσυνδεόμενα προκειμένου να αποφεύγετε το ενδεχόμενο να μην συνεργάζονται οι χώρες στις συμφωνίες ε, επιστροφής. Σε ό,τι αφορά τις ανθρωπιστικές ε, θεωρήσεις, ξέρετε ποια είναι η άποψή μου. Είναι το επόμενο θέμα αυτό στην ημερήσια διαταξή, αλλά συνδέεται με το θέμα μα. Σε ό,τι αφορά τι ανθρωπιστικέ λοιπόν θεωρήσει, τι θεωρήσει για ανθρωπιστικού λόγου, ε, πιστεύουμε ότι τα κράτη-μέλη ήδη έχουν ε, έκαστο ένα σύστημα για θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους και δεν μας φαίνεται σκόπιμο να παρέμβουμε στις εθνικές αρμοδιότητες, χορηγώντας τέτοιου είδους θεωρήσεις. Καλό θα ήταν η Ευρώπη να μείνει εκτός των θεωρήσεων αυτών. Να το αφήσει αυτό στα χέρια των κρατών μελών. Γιατί στη τελική ανάλυση τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία πρέπει να μπορούν να αποφασίσουν ποιο μπαίνει και ποιο δεν μπαίνει στην επικράτειά του. Γι' αυτό λοιπόν και συνεχίζουμε να αρνούμαστε την σύνδεση αυτή μεταξύ θεωρήσεων και θεωρήσεων για ανθρωπιστικούς λόγου. Ξέρετε ποια είναι τη θέση μα την έχω επαναλάβει πολλές φορές ε, και νομίζω ότι είναι σαφής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε, Στίβα, κύριε Στίβενς. Ο κύριος Δεπρέ. Ευχαριστώ και εγώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να χαιρετήσω τις προσπάθειές σας. Γνωρίζω πόσο δύσκολο ήταν αυτό το θέμα και αρχικά ήταν υπέρ της συμπερίληψης των ανθρωπιστικών θεωρήσεων στο, στο Γενική Έκθεση για τις Θεωρήσεις. Τελικά δεν τα καταφέρατε, γι' αυτό ήταν δύσκολο να το διεκπαιρεώσετε. Ε, είπαμε όμως παράλληλη συζήτηση του κώδικα θεωρήσεων ε, και το θέμα των θεωρήσεων για θεωροπιστικούς λόγους. Σας ευχαριστώ που λάβατε υπόψη και πολλές τροπολογίες μας. Σας ευχαριστώ θερμά και Ακριβώ ε, με πνεύμα συνεργασία καταθέσαμε τι τροπολογίε και ελπίζω να γίνουν δεκτέ και από άλλε αντιπροσωπείε. Θα σταθώ όμω σε κάποια σημεία τα οποία δεν άκουσα στην αρχική σας ε, ομιλία. Καταρχήν, θα θέλαμε τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα για όλους του ετούντε ε, να υποβάλουν απευθεία το αίτημά του στο προξενείο του, στο προξενείο μια χώρα μέλου. Δεν είμαστε κατά του παρόχου υπηρεσιών. Θεωρούμε όμως να, ε, ότι σκόπο είναι να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα. Δεν μας είπατε επίσης τίποτα για το εξή θέμα. Θέλουμε οι αιτήσει να γίνονται το νωρίτερο 9 μήνες πριν την έναρξη του ταξιδιού. Γιατί? Πολλές, ε, πολλά τέτοια ταξίδια γίνονται αεροπορικά και οι τιμές των εισιτηρίων ε, εξαρτώνται από το πότε θα τα αγοράσει κανείς. Αν θέλουμε λοιπόν να εθαρρύνουμε τον τουρισμό και να επιτρέψουμε σε οικογένειες να επισκεφθούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, θέλουμε να διαβριθεί αυτή η προθεσμία και όχι να, συντομευθεί. Σε ό,τι αφορά το τέλος θεώρησης. Εμείς ήμασταν υπέρ της αύξησης των τελών θεωρήσεων, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητούμε όμως τρεις διορθώσεις. Πρώτον, όταν κάποιος ζητά θεώρηση και ήδη υπάρχουν διαθέσιμα τα βιομετρικά του στοιχεία και μάλιστα είναι έγκυρα, να μπορεί να υποφελείται από μία μείωση. Γιατί τότε το κόστος όντως μειώνεται αισθητά. Θεωρούμε ότι το κόστος θα πρέπει να μειωθεί για τα παιδιά 6 έως 18 και τα μέλη της οικογένειας ενός υπηκότης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπει το άρθρο 5 της Οδηγίας του 2004-38, να μην καταβάλουν τέλη θεωρήσεων, γιατί το άρθρο 5 το προβλέπει ρητά. Σε ό,τι αφορά το, την προθεσμία επεξεργασία του αιτήματο. Θεωρούμε ότι η δεκαήμερη προθεσμία είναι λογική. Θα μπορούσε όμω να συντομευθεί για του αιτούντε θεώρηση όπου ήδη έχουν ε, τα βιομετρικά του στοιχεία εγγεγραμμένα στο σύστημα θεωρήσεων Σέγγεν. Σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση με την επανεισδοχή. Εσείς είστε επιφυλακτικός. Εμείς είμαστε υπέρ αυτού του συνδέσμου όμως με την επανεισδοχή και από ό,τι κατάλαβα είστε έτοιμος ε, να δεχτείτε την πρότασή μας, δηλαδή να μην ε, τιμωρούμε τους ε, πολίτες, αλλά τους ηθήνοντες των χωρών αφαιρώντας τους από τις διευκολύνσεις όταν αυτοί οι θύνοντες δεν δέχονται να συνδέσουν τις θεωρήσεις με την επανεισδοχή. Τέλος, ζητήσαμε και δεν το σχολιάσατε. Ένα χρόνο μετά τη θέση ίσχυ του κανονισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει έκθεση αξιολόγηση για την κατάργηση των βινιατών θεωρήσεων και τη θέσπιση μια ψηφιακή θεώρηση. Γιατί μπαίνουμε σε μια νέα εποχή, την ψηφιακή εποχή, με την ανάπτυξη νέων τεχνολογικών. Κρίνουμε λοιπόν σκόπιμο, κύριε Πρόεδρε, ε, σκόπιμο και ε, ευάρεστο να ζητούμε από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταθεί στο ύψος των τεχνολογικών εξελίξεων της εποχής μας, μια και υποτίθεται ότι ε, καυχάται για εξυγχρονισμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κυρίως για την καλή σας προσπάθεια και ε, επιμονή να ξεφύγουμε από το διέξοδο στο θέμα αυτό. κυρία Βεαχζιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να εκφράσω την ευχαρίστησή μου για την αγαστή μας συνεργασία. Και πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε συμφωνία, αρκεί να μην ε, κάνουμε τη διάκριση μεταξύ των εθεροβαμόμενων και αυτών που ε, μεριμνούν για την ασφάλεια των πολιτών. Νομίζω ότι όλοι ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια των πολιτών. Εδώ και χρόνια παρακολουθώ το θέμα των θεωρήσεων και είδα τις εξέλιξεις από την πρώτη μεταρρύθμιση του κώδικα θεωρήσεων. Θα ήθελα λοιπόν να συνεχίσουμε να σεβόμαστε ημέν μεν τους δε και ημέν μεν τις θέσεις των δε. Και μάλιστα το θέμα των θεωρήσεων δίνει μια εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο και με την πολιτική μας για τις θεωρήσεις δίνουμε κάποια στοιχεία στον υπόλοιπο κόσμο. Και θέλουμε να προσελκύσουμε επισκέπτες στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια στα πλαίσια του δικαίου της ελεύθερης διακίνησης και του σχετικού δικαιώματος. Αυτά που είπαμε για τους αθλητές, για τους καλλιτέχνες, για τους φοιτητές, για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ισχύουν. Προσοχή να μην ε, βλάψουμε ή να μην ε, πλήξουμε ανάλογα με τα μέσα που έχει ο καθένας ε, τη δυνατότητά του να ταξιδέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες πολιτών που αν δεν τους εξαιρέσουμε τουλάχιστον να απαλλάξουμε ανηλίκους κάτω των 18 ετών από, τα, την υποχρέωση τέλη καταβολής τελών θεωρήσεων. Και νομίζω τα 18 χρόνια είναι λογική ηλικία. Επίσης, ε, να προβλέψουμε δυνατότητα μείωσης ε, των τελών υπόρους. Όταν κάποιος είναι ε, ήδη εντεταγμένο στο σύστημα Σέγγεν για τις θεωρήσεις ή κάποιες άλλες κατηγορίες, νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε για μειώση των τελών σε κάποιες περιπτώσεις. Λυπάμαι και φαντάζομαι θα το περιμένατε ε, λυπάμαι που αποκλείσαμε τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις από το όλο θέμα. Πάντως, ε, για το αίτημα προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, που είτε μας αρέσει είτε όχι εμπίπτει στο θέμα των θεωρήσεων, γιατί τα κράτη-μέλη δέχονται αυτές τις πιθανότητες και εκεί ζητούμε ε, να υπάρχει αυτή η διάσταση, να ληφθεί υπόψη η ανθρωπιστική διάσταση σε αντίθεση με πολλούς συναδέλφους και κυρίως ε, σε αντίθεση με τους προλαλήσαντες, εμείς είμαστε κατά ε, της υπεργολαβίας τους παρέχοντες υπηρεσία, γιατί φοβόμαστε μήπως σε κάποιες χώρες ε, οδηγηθούμε σε καταχρήσεις με αυτή τη δυνατότητα εκχώρηση σε παρόχους υπηρεσιών. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε λοιπόν να περιορίσουμε αυτές τις καταχρήσεις. Συμφωνώ με τον κύριο Τεπρέ ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να αποκλείουν, αποκλείουμε οποιαδήποτε δυνατότητα υποβολής ε, του αιτήματο ε, στα προξενία ή στις πρεσβείες. Θα πρέπει να υπάρχει εναλλακτική. Σε καμία περίπτωση να μην είναι μοναδική λύση ή πάροχη υπηρεσιών. Είμαστε υπέρ του περιορισμού του κόστους ε, των παρόχων υπηρεσιών, γιατί γνωρίζουμε ότι γίνονται κάποιες καταχρήσεις εκεί. Επίσης, είμαστε υπέρ της επιστροφής των τελών θεωρήσεων για εκείνους που δεν ε, έγινε δεκτό το αίτημά τους, γιατί σε πολλές χώρες ε, οδηγούμαστε σε υπέρογκα ποσά που χρειάζεται να καταβάλουν κάποιοι που τελικά δεν έχουν καμία πιθανότητα να λάβουν θεώρηση. Η πολιτική θεώρηση δεν θα πρέπει να είναι πολιτική του κόστους και η επιλογή δεν θα πρέπει να γίνεται με βάση το κόστος. Και με το ίδιο πνεύμα θα θέλαμε οι οικογένειες να απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρηση για μερικέ περιπτώσει, ιδιαίτερα όταν συνοδεύουν παιδιά για κάποιε καλλιτεχνικέ ή αθλητικέ εκδηλώσει. Γιατί έχετε αυτή την αιμονή και δεν θέλετε να απαλλάσσουμε τι οικογένειε από την υποχρέωση θεώρηση, Νομίζω ότι αυτό είναι τμήμα του συνόλου. Και τέλο, σε ό,τι αφορά το σύνδεσμο με την επανεισδοχή. Γνωρίζετε ότι η ομάδα μα διαφωνεί με τη διασύνδεση τη κινητικότητα με την επανεισδοχή. Πάντως, η πρόταση του κυρίου Ντεπρέ είναι λογική. Γιατί αυτό που μας προβληματίζει κυρίως ε, είναι η υπήκοοι των τρίτων χωρών να μην γίνουν έρμεα όμοιροι των κυβερνήσεών τους. Γιατί δεν φταίνουν οι πολίτες για την πολιτική των κυβερνώντων τους και δεν θα πρέπει να στερούνται ε, οι πολίτες θεωρείς, αλλά οι θύνοντες, οι κυβερνώντες. Ιδιαίτερα για τις χώρες που υπάρχει ανάγκη θεώρησης για ανθρωπιστικούς λόγους. Και εκεί θα ήταν επικίνδυνο οι χώρες ε, που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, να, οι πολίτες να μην έχουν δικαίωμα να ζητήσουν θεώρηση. Γιατί έτσι πλήττονται διπλά. Είμαι πάντως ε, έτοιμη να συνεργαστώ για να καταλήξουμε συμβαστικές λύσεις για πάρα πολλά σημεία και γιατί όχι και σε όλα τα εκκρεμή σημεία. Ευχαριστούμε κυρία Βερζιά. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ όλους θερμότατα για τα σχόλιά σας και επιμένω ότι είναι προφανές και εγώ ως συγητής έκανα ό,τι μπορούσα, έβαλα τα δυνατά μου και χάρη στη δική σας συνεργασία ε, προχωρήσαμε. Ζητώ λοιπόν να κάνετε αυτή την ίστατη προσπάθεια για να καταλήξουμε σε λογικές συμβαστικέ λύσεις. Με ακούσατε επανειλημμένος ε, να λέω με πόνο καρδία ότι πλησιάζουμε στο τέλος κοινοβουλευτική θητείας. Και με προβληματίζει ιδιαίτερα η, η δράση της Επιτροπής και τα αποτελέσματα των εργασιών μας γιατί είμαστε Επιτροπή Πολιτικών ε, Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών. Θα πρέπει λοιπόν να προσφέρουμε έργο, να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Έτσι θα δείξουμε την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε στις ανησυχίες των συμπολιτών μας. Γι' αυτό και σας θέρμο παρακαλώ να κάνουμε όλοι μια ίστατη προσπάθεια, να συγκλίνουμε τις απόψεις μας και να καταλήξουμε σε εφικτές και λογικές συμβαστικές λύσεις. Κατέγραψα προσεκτικά όλα σας τα σχόλια και είμαι έτοιμος να κάνω και εγώ αυτό το τελευταίο βήμα. Και μάλιστα έχουμε προγραμματίσει την Τετάρτη τεχνική συνεδρίαση στις 12 το μεσημέρι. Τετάρτη 12 το μεσημέρι τεχνική συνεδρίαση για να κάνουμε όλη αυτή την ίστατη προσπάθεια και να καταλήξουμε στις συμβαστικές λύσεις. Και σας διαβεβαιώ για να κερδίσουμε και χρόνο, γιατί μας ε, πιέζει και ο χρόνος και τα το γεμάτο πρόγραμμα που έχει συνήθως η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, είμαστε υποχρεωμένοι να συνοψίσουμε όσο γίνεται τα θέματα και να καταλήξουμε σε περιληπτικές συμβαστικές τροπολογίες. Πάντως λάβω υπόψη πολλά στοιχεία σα, Για παράδειγμα, δυνατότητα έκδοσης θεωρήσεων σε προξενία και πρεσβείες. Να μην χρειάζεται κανείς να προσφεύγει σε εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών. Επίσης, σημείωσα αυτό που είπατε για την αξιολόγηση που θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Με μια έκθεση που θα αντλεί διδάγματα από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας από την εφαρμογή του συστήματος θεωρήσεων. Επίσης, ε, σημείωσα τα σχόλια του κυρίου Ντεπρέ και μάλιστα πολλά από αυτά ήδη έχουν λεφθεί υπόψη στην έκθεσή μου. Φυσικά και η δυνατότητα μείωση των τελών το θεωρήσω για όσους έχουν ήδη ε, μετέχουν στην τελευταία εκδοχή του ΒΙΣ, του συστήματος θεωρήσεων Σέγγεν. Θα κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε, θα βάλουμε τα δυνατά μας και κάνουμε μια ίστατη προσπάθεια για να καταλήξουμε σε συμβασμούς. Σας παρακαλώ συνεργαστούμε για να έχουμε αποτελέσματα, γιατί αλλιώς δεν θα είναι ικανοποιητική η θητεία μας. Και μια και πλησιάζουμε στο τέλος της συνεδρίασης, να κάνω κάποια σύντομα σχόλια για τη συμπληρωματική μου έκθεση, που επίσης είναι έκθεση πρωτοβουλίας για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις. Ε, μου είναι ιδιαίτερα προσφυλής. Γνωρίζετε την κατάσταση. Η διάσκεψη των Προέδρων έκανε μία πρόταση να δοθεί άδεια στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, να υποβάλει νέα έκθεση πρωτοβουλίας για να ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου με το ίδιο θέμα. Γιατί είδατε τι διαμαρτυρίες υπήρξαν για δυσαρέσκειες με την τελική έκβαση και κυρίως για το γεγονός ότι η τελική έκβαση εξαρτώνταν από το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη είχαν ήδη αποσύρει ε, την ε, έγκρισή τους κατά την φάση, τελική φάση του ελέγχου. Πρόταση είναι να υιοθετηθεί με τη συνοπτική διαδικασία, τη διαδικασία fast track έκθεση, ώστε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Οπότε, σας έχουμε ήδη μοιράσει πριν τη συνεδρίαση το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε το ίδιο επιτελείο, την ίδια ομάδα, τον ίδιο συγγητή, τον υποφαινόμενο, του ίδιου και οδησυγητές ε, που ορίστηκαν από τους συντονιστές της ΛΥΜΠΕ. Και γι' αυτό η προθεσμία θα είναι όσο το δυνατό πιο σύντομη γίνεται. Είναι σχεδόν τυπική αυτή η προθεσμία. Μια και δεν θα πρέπει να αμφισβητηθεί η πολιτική συμφωνία, ούτε να ξανανοίξουμε συζήτηση για κάποια θέματα. Θα πρέπει να εμείνουμε στο κείμενο που είναι η απόρρια των διαπραγματεύσεων και μόνο έτσι θα έχουμε έτοιμο κείμενο για ψήφο στη ΛΥΜΠΕ 3 Δεκεμβρίου και τελική ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου, στο Στρασβούργο. Προσπαθώ να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα για την Τρίτη Τετάρτη στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου και πιστεύω ότι είναι λογικό γιατί Δευτέρα δεν έχουν έρθει ακόμη όλοι και την Πέμπτη ήδη έχουν φύγει μερικοί στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, οπότε θα φροντίσω να μπει να προγραμματιστεί η ψηφοφορία για την Τρίτη Τετάρτη στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατό πιο περισσότερες θετικέ ψήφους γίνεται. Σας υπενθυμίζω ότι χρειαζόμαστε ενισχυμένη πλειοψηφία για τις ανθρωπιστικές θεωρήσεις, ώστε να για να βρούμε λοιπόν την ισορροπία αυτών των διαφόρων θεμάτων και για να προλιάνουμε το έδαφος για συμφωνία. Ζητώ και πάλι τη συνεργασία σας και τη στήριξή σας, ώστε να εμείνουμε στο αρχικό κείμενο της Ολομέλης, γιατί τίποτα δεν έχει αλλάξει στο μεταξύ. Ουσιαστικά υποβάλλουμε το ίδιο κείμενο που ήταν το αποτέλεσμα συμφωνίας των πολιτικών ομάδων και είχε υπερψηφιστεί στο παρελθόν στη Λίμπε. Για να είμαστε λοιπόν συνεπεί και συνεκτικοί και να στείλουμε το σωστό μήνυμα στους Ευρωπαίους πολίτε και στην κοινή γνώμη που έχει στραμμένα τα μάτια της πάνω μας και περιμένει μια απάντηση από εμά στο συγκεκριμένο θέμα, σα ζητώ και πάλι να επιδείξετε συνεργατικό πνεύμα για να μπορέσουμε να διεκπαιρεώσουμε αυτό το θέμα των ανθρωπιστικών θεωρήσεων και να ψηφίσουμε στις 3 Δεκεμβρίου στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και στις 10 ή 11 ή 12 Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια του Στρασβούργου. Ας συνεργαστούμε παρακαλώ για να τα καταφέρουμε. Ποιος θέλει το λόγο, η κυρία Γκόμες που σήκωσε το χέρι από ό,τι είδα. Πρόεδρε, να σας υποστηρίξω, να σας υποστηρίξω απόλυτα. Και να απευθύνω κι εγώ έκκληση να υποστηριχθεί η γραμμή την οποία προτείνεται ως μέλος του Κοινοβουλίου. Πραγματικά αισθάνεται φρικτά. Μετά από αυτά που είδα στην τελευταία ολομέλεια, μας συμβαίνουν με την έκθεση αυτή. Ελπίζω να ήταν μια άτυχη στιγμή και όχι μια πολιτική τοποθέτηση των μεγάλων πολιτικών ομάδων στο Κοινοβουλίο. Σα υποστηρίζω. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπέκερ, παρακαλώ μου σύντομα, γιατί οι διερμηνεί μας θα πρέπει να φύγουν σε δύο λεπτά. Να είμαι σύντομο λοιπόν. Χαίρομαι καταρχάς που είχαμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε εκ νέου την έκθεση αυτή. Κάποιοι είχαν ψηφίσει πριν από την έκθεση και μετά δεν ψήφισαν την ανθρωπιστική θεώρηση. Ήταν ε, ίδιος αριθμός των σοσιαλδημοκρατών με εκπροσώπους ε, του ΕΛΚ. Άρα δεν υπάρχει κανένας ε, Λόγω να δημιουργούμε ιστορίε για το πολιτικό υπόβαθρο που υπάρχει. Δεν υπήρχε. Δεν ε, υπήρχαν ομάδε που ήταν κατά της έκθεση. Να ξεκαθαρίσω ότι στην παρούσα φάση δεν πιστεύουμε ότι κάποια στοιχεία είναι ξεκάθαρα διτυπωμένα. Θα υποβάλουμε διευκρινιστικές τροπολογίες προς τον εισηγητή Υπάρχουν συμβαστικές προτάσεις και από τον κύριο Ντεπρέ που θεωρούμε ότι δεν επαρκούν για να ξεκαθαρίσουμε ότι υφίστανται σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες των προξενείων και των πρεσβειών Δεν είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η θεώρηση για τους ανθρωπιστικούς λόγους ε, είναι κάτι το οποίο δεν υποστηρίζουν πολλοί συνάδελφοι. Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα υποστηρίξουν πιο πολλοί συνάδελφοι, λοιπόν. Θα ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά μια και δεν έχουμε χρόνο, να σας πω ότι κάποια θέματα εξακολουθούν να είναι ασαφή. Έχουμε χρόνο όμως να βρούμε συμβιβασμούς από κοινού. Ευχαριστώ. Η κυρία Βρισιά, θέλετε να πάρετε το λόγο. Ναι. Θα ήθελα να σας διευκρινίσω ότι η συνεργασία αυτή σε αυτό το επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι κάτι το οποίο ε, αποτελεί ευρωπαϊκό επίτευγμα. Είναι φυσιολογικό να θέλουμε να διαπιστώσουμε τι συνέβη και να μην αμφισβητείται η πλειοψηφία που πρέπει να υποστηρίξει το κείμενο Σα ε, Υπενθυμίζω ότι είναι ειδική πλειοψηφία, ειδική πλειοψηφία που ζητείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 349 ψήφους υπέρ και λιγότερες κατά. Νομίζω ότι η συμφωνία που επετέφθη στην διάσκεψη των Προέδρων για την κατάθεση του ίδιου κειμένου στα πλαίσια της ταχεία διαδικασία είναι σαφή. Δεν θέλουμε να ξανανοίξουμε το κουτί τη Πανδώρα. Δεν είναι η στιγμή να ξεκινήσουμε πάλι με του συμβιβασμού. Έχουμε το κείμενο ξεκάθαρα μπροστά μα και θα πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστώ. Μία τελευταία φράση. Είδατε τι έγινε. 26 άτομα, 26 ψήφοι μα έλειπαν για ειδική πλειοψηφία. Χρειαζόταν ειδική πλειοψηφία. Αυτό είναι το σωστό μήνυμα θα ήταν ε, αδύνατο να κατανοήσουμε αποτυχία του Κοινοβουλίου να αποστείλει ένα μήνυμα για την έκθεση αυτή. Αυτό περιλαμβάνει αρκετά σημεία για να περάσει με την ειδική πλειοψηφία στις πολιτικές ομάδες. Όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία προτάθηκαν μέσω των μακρών διαπραγματεύσεων έχουν ε, συνδυαστεί, έχουν ε, διατυπωθεί εγγράφος. Σας καλώ να κάνετε ό,τι μπορείτε για να διαβιβάσετε το μήνυμα αυτό προς τις πολιτικές ομάδες που προσωπείτε, προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι στην ψηφοφορία αυτή το Δεκέμβριο θα πετύχουμε το σκοπό μας. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό μήνυμα θα ήταν πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε μια αποτυχία. Σας ευχαριστώ και σας παρακαλώ λοιπόν να προσπαθήσετε να το πετύχουμε αυτό. And that's it, that, we're coming to the end of this afternoon session. Of course, we're resuming our works tomorrow by 9. Ολοκληρώσαμε την απογευματινή μας συνεδρία. Ραντεβού αύριο στις 9. Καλό σας βράδυ.